Ehm, Καλώς σας απόγευμα σε όλους. Ε, χαιρετίζω και όλους τους επισκέπτες που είναι στην Επιτροπή μας. έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό, που κάθε φορά γίνεται και πιο δύσκολο. Έχουμε δύο εισηγητέ, τον κύριο Ριβελίνη και την κυρία συγγνώμη, Γκρέσλε, που είναι εισηγητέ για το θέμα αυτό, των δημοσιονομικών κανονισμών που εφαρμόζονται στον προπολογισμό τη Ένωση. Και ω δείγμα του ενδιαφέροντο έχω αυτή τη στιγμή περίπου 500 τροπολογίε ως ε, αντιπρόεδρος της Προεδρεύω αυτής της Επιτροπής. Ξέρετε ότι ο κύριος Δεμαγίστρης έγινε δήμαρχος της Νάπολης και δεν έχει αντικατασταθεί ακόμα, επομένως πρέπει προς το παρόν τον αντικαθιστά κάποιος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Θα δώσω λοιπόν καταρχήν το λόγο στους εισηγητές και στη συνέχεια θα περιμένουμε να ακούσουμε τις, αν... τις αντιδράσεις των συνοδέλφων και θα δώσουμε μετά το λόγο στην ε, Κομισιόν. Ποιος από τους δύο συγγητές θα ήθελε πρώτος να λάβει το λόγο. Ο κύριος Ριβελίνη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λαμβάνω το λόγο λοιπόν για το δημοσιονομικό κανονισμό και εδώ θα πρέπει να διευκρινίσω ότι έχουν κατατεθεί άλλες 260 τροπολογίες που προστίθενται στις 220 τροπολογίες που είχε η προηγούμενη που είχε η έκθεσή μας όταν παρουσιάστηκε από τους δύο συνεισηγητές. Είναι φανερό ότι πρόκειται για ένα θέμα μεγάλης πολυπλοκότητος. Είναι πολλά τα θέματα που προσπαθούν να τροποποιήσουν οι τροπολογίες ώστε να τροποποιηθεί ο τρέχον δημοσιονομικός κανονισμός μεταξύ όλων αυτών. Είναι χρήσιμο να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει μια τροποποίηση του νομικού πλαισίου, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, που στο μέλλον θα έχει τη κανονισμού και επίσης το γεγονός ότι η διαθεσμική συμφωνία σε σχέση με την πειθαρχία του προϋπολογισμού και την χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση θα ενσωματωθεί μέσα στον ίδιο αυτό τον κανονισμό. Έχουμε λοιπόν την ε, επέκταση της αρχής ότι μόνο για τον επόμενο χρόνο θα μπορούν να μεταφέρονται οι υποχρεώσεις που έχουν ε, συναυθεί μόνο μία φορά θα μπορούν να μεταφερθούν, μόνο στον επόμενο χρόνο. Ακόμα και σε περίπτωση πλήρους μη χρησιμοποίησής τους. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να υπάρξει ένα γενικό πλαίσιο στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να δημιουργηθεί επίσης ένα σύστημα προστασίας κατά των ε, ατασταλιών και απατών που εξασφαλίζει και την κάλυψη του κόστους των συστημάτων ε, ελέγχου του προϋπολογισμού. αυτές είναι ανθρωπολογίες 270 και επέκεινα, η δημιουργία ενός επίσης σαφούς συστήματος που να περιλαμβάνει το κόστος προσωπικού για τα θέματα αυτά, είναι τροπολογία 300 και στη συνέχεια έχουμε διευκρινίσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η από κοινού διαχείριση, ποιε θα πρέπει να είναι οι ευθύνε των κρατών μελών και ιδίω την ανάγκη η δράση των κρατών μελών να έχει σαν στόχο την προάσπιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ελέγχους και εξάντε και εξπόστ. Αυτές λοιπόν είναι οι καινοτομίε οι οποίες τίθενται. Ξέρουμε όμως ότι οι επόμενοι μήνες δεν θα είναι εύκολοι. Ε, θα έχουμε μια μακρά και δύσκολη συζήτηση με το Συμβούλιο η οποία θα πρέπει να περατωθεί ιδίως για το άρθρο 66 που αφορά τα συστήματα ε, διαπίστευσης και τις ε, προϋποθέσεις για την αναστολή των πληρωμών. Πριν κλείσω λοιπόν την παρέμβασή μου και αφήσω το λόγο στην κυρία Γκρέσλε, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση και να υποβάλω μια πρόταση ή διευκρίνηση. Είδα ότι πολλοί συνάδελφοι παρουσίασαν τροπολογίες για το άρθρο 29 που κινούνται προς την κατεύθυνση της διαγραφής της έννοιας ενός αποδεκτού περιθωρίου σφάλματος. Ενώπιον αυτών των τροπολογιών, εγώ θέλω να υπενθυμίσω στους συναδέλφους για το γεγονός ότι εμείς ως εισηγητές προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Κομισιόν, η οποία είχε ε, εντοπίσει αυτή την έννοια του ε, ανεκτού περιθωρίου σφάλματος για, να, για, τις, για τους ελέγχους και μόνο. η πρότασή μας κατόπιν υπόδειξης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εισάγει μια έννοια νέα για τον ανεκτό κίνδυνο που ενεργοποιείται όχι μόνο από το κράτος μέλος αλλά και από τα ταμεία και γίνεται ένα ε, σύστημα ένα εργαλείο διαχείρισης. Θα ήθελα να σας κάνω έκκληση να σκεφτείτε ότι η εισαγωγή αυτού του εργαλείου όπως προτείνεται δεν θα τροποποιήσει το κατόφλι του 2% στη μεθοδολογία εργασίας του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα δημιουργήσει ένα επίπεδο κινδύνου ανεκτό και έτσι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα εξηγήσουν αλλά ότι και η παραμικρή ε, υπέρβαση θα είναι απαράδεκτη. Επίσης, σε τομείς που υπάρχει λάθος πάνω από 5% βρισκόμαστε στην λεγόμενη κόκκινη ζώνη. Και αν περάσει η σχετική μας τροπολογία, αυτό δεν θα ξανασυμβεί στο μέλλον. Το λέμε, αυτό στην Κομισιόν το ξέρει. Επίσης, θέλω να σας πω ότι υπάρχει και μια προφορική τροπολογία που θα μπορούσε να, τη χρησιμοποιήσουμε για να επιλύσει το πρόβλημα για την απαλλαγή των υπολείπων θεσμικών οργάνων ε, πέρα από την Κομισιόν για τις οποίες ήμουνα ε, εισηγητής. Με αυτόν τον τρόπο η εμπειρία που είχα ως ε, εισηγητής θα προσπαθήσει να βρει μια λύση Διαρκεί για το πρόβλημα όλων των απαλλαγών, όλων των θεσμικών οργάνων. Νομίζω ότι η Γραμματεία ε, μοίρασε το κείμενο το οποίο θα σας διαβάσω. Άρθρο 156. Μιλάμε για τη διαδικασία της ε, απαλλαγής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, κατόπιν ε, συμβουλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Συμβουλίου, συγγνώμη, με ειδική πλειοψηφία μέχρι το, τις 15 Απριλίου του χρόνου νησιν 2 δίνει απαλλαγή ε, για την τρέχουσα χρονιά. Εν συνεχεία, έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε τις άλλες, τα άλλα θεσμικά όργανα, ε, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1-2 και τα, τις υπόλοιπες οντότητες που αναφέρονται στο 196 β παράγραφος 1 και άλλοι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των κοινοτικών ταμείων ε, σε ό,τι αφορά την διαδικασία της απαλλαγής για, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως προβλέπεται από την κοινωνική, κοινοτική νομοθεσία. Και τώρα το λόγο έχει η συνάδελφος. Ευχαριστώ. Το θέμα αυτό όλοι το λένε σημαντικό και κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί. Γι' αυτό ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Δύο έγγραφα φέραμε. Το ένα είναι καινούριο έγγραφο εργασίας. Ασχολούμεθα με τις τροπολογίες και την κριτική ε, της Κομισιόν. Το άλλο είναι έγγραφο της Γραμματείας. Ευχαριστούμε πολύ. Όπου η Γραμματεία μας λέει ποιε ποιες τροπολογίες κατατέθηκαν σε ποια άρθρα. Βλέπετε εδώ ένα σκιαγράφημα. Σε όλους αρέσουν αυτά οι εικόνες. Πάνω σε αυτή την εικόνα θα μιλήσω σήμερα. Έτσι έχουν τα πράγματα στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Αυτός ε, ο πίνακας ε, συμπεριλήφθη σε μια μελέτη μετά από έτοιμά μας. Είναι μελέτη από την Deloitte δημοσιονομικοί κανόνες, ε, ε, κανόνες εξυγχρονισμού για τα προγράμματα έρευνας. Αυτά είναι μια έρευνα που έγινε μετά από ανάθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμού πριν από λίγα χρόνια, υπό μου μετά από δική μου πρόταση. Το έχετε όλοι, επάνω έχετε τις συμβάσεις, μετά έχουμε το δημοσιονομικό κανονισμό και εφαρμοστικοί κανόνες που είναι ουσιαστικά η κατεξουσιοδότηση πράξης. Εφιστώ την προσοχή σας αυτά εδώ που είναι η κατεξουσιοδότηση πράξης. Βλέπετε πόσο ογκώδες είναι το κείμενο. Από αυτές τις πράξεις κατεξουσιοδότηση, γνωρίζοντας την ποικιλία των κανόνων, είναι 272 άρθρα, έχουμε καταλήξει σε αυτό εδώ το ε, έγγραφο, δηλαδή από τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, ε, αυτά θα τα κάνει η Κομισιόν, αυτά τα βγάλαμε εμείς, συνεχίζει η Κομισιόν με τα πολλά. Εμείς ε, επιλέξαμε αυτά γιατί εδώ έχουμε ουσιώδεις διατάξεις που συμπεριελάβαμε στο δημοσιονομικό κανονισμό για να αποφύγουμε τη μεγάλη καταστροφή των ενωσιακών κονδυλίων. Αυτό είναι το status quo εδώ δηλαδή επικαλυπτόμενοι κανόνες. Διαπιστώσαμε ότι εκεί όπου ο δημοσιονομικός κανονισμός δεν έχει κανόνες, ε, τότε οι κάτω βαθμίδες φτιάχνουν δικούς τους κανόνες. Έχουμε εδώ ας πούμε της κατεξουσιοδότηση πράξης, εδώ. Έχουμε τους κανόνες συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανόνες αυτοί. Μετά έχουμε το ίδιο το πρόγραμμα πλαίσιο, κανόνες ε, συμμετοχής για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρατόμ, δύο σειρές, τις βλέπετε εδώ. Αυτό που είναι το SP, τα SP είναι τα εξειδικευμένα προγράμματα μέσα στο πρόγραμμα για την έρευνα, το πρόγραμμα πλαίσιο, Marie Curie, έχουν διάφορα ονόματα, τα εξειδικευμένα προγράμματα και αυτά τα προγράμματα στα πλαίσια του προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα υπόκεινται σε δικούς τους κανόνες πάλι, κανόνες συμμετοχής. Υπάρχουν γενικοί κανόνες συμμετοχής που δεν συμπεριλαμβάνονται εδώ, εξειδικευμένοι κανόνες συμμετοχής, μετά ε, όταν διαπραγματεύτηκαν την ε, σύμβαση υπάρχουν και ε, συμφωνίες για τις επιδοτήσεις μεταξύ Κομισιών και τους δικαιούχους με το, και στο πρόγραμμα πλαίσιο και στα εξειδικευμένα προγράμματα υπάρχουν ε, κανόνες για την επιδότηση. Έχουμε και άλλους μέσα στα πλαίσια τα εξειδικευμένα, τα προγράμματα και εδώ σε αυτό το κομμάτι έχουμε το, μικρό, το G αυτό που είναι οι 20 κατευθυντήριες γραμμές μέσα σε 6 γενικές διευθύνσεις της ε, Κομισιόν που διαχειρίζονται κονδύλια για την έρευνα. Ε, μπορεί, μπορεί να είναι περίπου, περίπου σαν αυτό, λίγο λιγότερο, ε, οι 20 κατευθυντήριες γραμμές και αυτές πρέπει να τις ακολουθήσει όλες ο άμυρος ο δικαιούχος. Τι κρίμα, τον λυπούμεθα όλοι. Και επειδή τον λυπούμεθα, είπαμε να, δεχ, να εγκρίνουμε 20 άρθρα στο δημοσιονομικό κανονισμό από τους εφαρμοστικού κανόνες, ούτω ώστε να, μην, να το απογορεύσουμε αυτό το πράγμα να κάνει ο καθένας του κανόνες του. Έχουμε ας πούμε την εισφορά εισίδος, έχουμε τις επιδοτήσεις, ε, τις ε, δημοσιονομικές διορθώσεις, σημαντικά πράγματα. Αυτά που θεωρήσαμε ε, σημαντικά τα βγάλαμε από τους εξειδικευμένους κανόνες με την κρυφή ελπίδα ότι έτσι αυτή η πυραμίδα θα καταργηθεί. Θέλουμε να ε, ε, εναρμονίσουμε τους κανόνες. Βέβαια, εν μέρη, αντιφάσκουν μεταξύ τους οι κανόνες. Ε, γιατί χρειάζονται άνθρωποι να μας ερμηνεύσουν τους κανόνες. Πρέπει να φωνάξουμε ανθρώπους να μας πούν τι θα κάνουμε με τους, όλους αυτούς τους κανόνες. Αυτό είναι που θέλουμε να αποφύγουμε. Θα ξεκαθαρίσουμε πράγματα άπαξ και διαπαντός. Όπως ας πούμε ε, πώς θα υπολογίζομαι κατά αποκοπήν ποσά χρηματοδότησης. Αυτά είναι πολύ τεχνικά θέματα τα οποία προσπαθήσαμε να τα ρυθμίσουμε με τους δικαιούχους, με τις ενώσεις τους. Προσπαθήσαμε σε συμφωνία με τους ε, ενδιαφερομένους να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και με την Κομισιόν ε, και με τους ενδιαφερομένους πώς θα γίνουν σωστά τα πράγματα. Η εναρμόνιση των κανόνων τι σημαίνει ότι όλα αυτά θα τα ε, αναδιαρθρώσουμε για να καταλήξουμε σε καλύτερα αποτελέσματα και να μην αφήνουμε αμφιβολίες ερμηνείας. Έχουμε πολλά ερωτηματικά η Κομισιόν λέει ότι είναι γραφειοκρατικά αυτά που λέμε. Άμα είναι αυτά γραφειοκρατικά, τι είναι αυτή η πυραμίδα. Εγώ συμβουλεύω να συμφωνήσετε μαζί μας γιατί άλλη ε, διέξοδος δεν υπάρχει. Όλο αυτό το ε, όλη αυτή η υπόθεση θέλουμε να λήξει ειρηνικά και νομίζουμε ότι θα καταφέρουμε να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν υπάρχει ε, εύλογη εναλλακτική από αυτήν για να ε, εκτελεστεί ο προϋπολογισμός και σε ορισμένους ε, προαιρετικούς κανόνες να ε, έχουμε ενιαία ερμηνεία και ενιαία υλοποίηση. Τώρα δίνουμε μάχη με τη γραμματεία και ευχαριστούμε τη γραμματεία και από τον προϋπολογισμό και από τον έλεγχο προϋπολογισμού τους υπεύθυνους των γραμματιών γιατί μας βοήθησαν να βρούμε έναν τρόπο να βρούμε και να προτείνουμε συμβιβαστικέ λύσεις. Αν δείτε την πρόταση, το κείμενο της γραμματείας για τον αριθμό των τροπολογιών, ε, βλέπουμε ιδιαίτερα το άρθρο 56 να παίζει ρόλο. Έχουμε περίπου 70 ε, για ε, για την επιμερισμένη διαχείριση και ελπίζουμε ότι του θα κάνουμε μια καινούργια συμβιβαστική πρόταση που θα προσπαθήσουμε να τη συζητήσουμε με όλους. Γιατί αυτό έτσι όπως είναι είναι ε, take it or leave it. Ε, πιστεύουμε ότι πρέπει λειτουργικά, ε, να είναι λειτουργική η πρόταση. Δεν έχει νόημο να λειτουργήσουμε εμβαλωματικά και να παίρνουμε ένα στοιχείο από εδώ και ένα από εκεί αποσπασματικά. Θέλουμε να, κάτι που να έχει νόημα σε ό,τι αφορά τους όρους ας πούμε πιστοποίησης ε, για τα, στα κράτη-μέλη θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας για να διαμορφώσουμε κάποιες προτάσεις. Ο συνάδελφος Γκάιερ ρώτησε ε, ότι ποια εναλλακτική, ε, ποια είναι αυτή η καινούργια εναλλακτική για το άρθρο 56 ή η τρίτη ή η τέταρτη. Εν πάση περιπτώσει πρέπει κάπου να καταλήξουμε, δεν γίνεται αλλιώ. Σας παρακαλώ να αντισταθείτε στο λόμπινγκ της Κομισιόν. Επίσης χρειάζεται μια διαπραγματευτική θέση ε, και απέναντι στην Κομισιόν ε, το ε, Συμβούλιο δεν είναι χοροδία της περίκη χοροδία. Ξέρουν, είναι άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν συγκεκριμένους στόχους. Εάν θέλουμε και εμείς να κάνουμε κάτι και στο θέμα της απαλλαγής που ανέφερε ο κ. Ζιβελίνη και όταν θέλουμε να ε, έχουμε αποτελέσματα, κάτι πρέπει να προτείνουμε και να έχουμε διαπραγματευτική θέση συγκεκριμένη. Έμενα μου είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, της επιχείρη, το επιχείρημα ότι γραφειοκρατιοκοπιούμε την κατάσταση, αυτό να το καταρρύψουμε, γιατί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ε, είναι το αντίθετο από αυτό που ισχύει, γιατί τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τους δικαιούχους. Εμείς εξετάσαμε, αφού παρακολουθήσαμε επί χρόνια την κατάσταση, παρουσιάσαμε μια πολύ ενδελεχή ανάλυση τι ακριβώς συμβαίνει. Ε, στείλαμε την Πέμπτη μια επιστολή στους συναδέλφους όπου εκφράζουμε αυτή την ανάγκη εναρμόνισης των κανόνων. Σήμερα έχουμε το νέο έγγραφο εργασίας όπου καταπιανόμαστε με την κριτική της Κομισιόν και εξηγούμε πάλι τις τροπολογίες μας και θα το ξανακάνουμε αυτό γιατί αυτή είναι μια συνεχιζόμενη εργασία. Εν πάση περιπτώσει θα έχουμε μια κοινοβουλευτική θέση η οποία θα διαφυλάσει κατά στο μέγιστο βαθμό τα δικαιώματά μας αλλά θα ανταποκρίνεται και στη συνθήκη της Λισαβόνας με τους νέους κανόνες που μπορούμε να κάνουμε εμείς και, το, και τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν. Αυτά θα πρέπει να είναι διακριτά. Ό,τι δεν καταφέρνουμε δεν θα τα καταφέρουμε τα επόμενα 20 χρόνια. Δεν θα ξανάρθει δηλαδή αυτή η ε, καλή στιγμή. Ό,τι δεν περάσει τώρα θα το έχουμε χάσει για πολλά χρόνια. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ τους εισηγητές, την κυρία Γκρέσλερ που λέει ότι το Συμβούλιο δεν είναι παιδική χοροδία όντως Αλλά πρόκειται για μάχη που πρέπει να δώσουμε το Συμβούλιο εμείς στο Κοινοβούλιο και θα πρέπει να επιβληθούμε. Λοιπόν, θα πρέπει να διαχειριστούμε λίγο το χρόνο. Έχουμε 30 λεπτά για να ακούσουμε τους συναδέλφους. Θα δώσουμε το λόγο και στην Κομισιόν βέβαια. Υπάρχουν διάφοροι συνάδελφοι που φτάσαν τώρα. Ποιο θα ήθελε παρακαλώ να πάρει το λόγο, να δω πόσοι θέλουν το λόγο καταρχήν. Ποιοι θέλουν να πάρουν το λόγο σε αυτή τη συζήτηση, παρακαλώ μετά από την παρουσίαση των δύο εισηγητών. Κανείς, ουδής. Κανείς άλλος. Ο κύριος Μιούλερ. Και ο κύριος Οντί. Ο κύριος Μιούλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ανάλυσα τις διάφορες τροπολογίες και έπαθα πάνω κέφαλο. Άρχισα να μου γυρνάει το κεφάλι γύρω-γύρω. Μου άρεσε αυτή η σύγκριση που κάνατε με τη ζυγαριά και τα λοιπά στις τροπολογίες. Αλλά αν εκτελέσουμε όλες τις τροπολογίες, αν περάσουμε στις τροπολογίες, η κατάσταση θα περιπλακεί, μου φαίνεται πολύ περισσότερο. Θα ήθελα λοιπόν οι εισηγητέ να μα παρουσιάσουν συμβαστικέ τροπολογίε στο συντομότερο δυνατό. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο. Ανέλησα μια σειρά από τροπολογίες, ασχολήθηκα με τους διάφορους ε, παράγοντες κινδύνου και η πρόταση νομίζω τη κύρια Γκρέσλα είναι θαυμάσια. Αλλά υπάρχουν και διάφορες άλλες προτάσει. Καλό θα ήταν να αναλύσουμε τους συμβιβασμούς, να τους αναλύσουν οι εισηγητές δηλαδή. Συγγνώμη, να αναλύσουμε εμείς τους ε, συμβιβασμούς των εισηγητών και να ακούσουμε και κανένα σχόλιο από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι άποψη έχει. Το Συμβούλιο θα πάρει και αυτό το λόγο αργότερα, αλλά να μου πει η Κομισιόν τι είναι υλοποιήσιμο και τι όχι. Γιατί ε, βλέπω συνέχεια να υπάρχει όρος πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Ε, πράξεις κατά ανάθεση, ανατιθέμενες πράξεις. Ε, το ακούω υπό όλες τις ε, μορφές του λόγου. Θέλω να καταλάβω περί τίνος πρόκειται ακριβώς. Θα ήθελα λοιπόν μια απάντηση της Κομισιόν. Αυτή η αναθεώρηση, γιατί έχω δει πολλούς, πολλές αναθεωρήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού, δεν είμαι φρέσκος εδώ, ε, γιατί αυτή η αναθεώρηση είναι μοναδική ευκαιρία. Ε, και αν, εν πάση περιπτώσει, σε τρία χρόνια δούμε ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος, γιατί δεν θα μπορούσαμε δηλαδή να αναθεωρήσουμε και να διορθώσουμε αυτόν τον κανονισμό. Οι, οι λοιπόν, θα ήθελα να κάνουν συμβαστικές τροπολογίες και περιμένω και την αντίδραση της Κομισιόν. Ο κύριος Σοντή τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ουσιαστικά θέλω να πάρω το λόγο για δύο θέματα. Θέλω καταρχάς να συγχαρώ τους δύο συγγητές που κάνουν μια δύσκολη αλλά απαραίτητη δουλειά. Έχω καταθέσει μια σειρά από τροπολογίε για το χρονοδιάγραμμα των απαλλαγών, της απαλλαγής. Προτείνω λοιπόν να κλείσουμε τη διαδικασία απαλλαγής την επόμενη χρονιά ε, από αυτή που ελέγχουμε. Όταν συζητώ με άλλους ευρωβουλευτές, ειδικού ή όχι, τους φαίνεται λογική αυτή η πρόταση. Συζητώντας όμως με τους πραγματικά ενδιαφερόμενους, την Κομισιόν, τα μέλη του δικαστηρίου κτλ. Μου λένε ότι υπάρχουν πολλά τεχνικά προβλήματα με αυτή την πρόταση. Θέλω να πω στους ηγητές μας λοιπόν ότι εγώ δεν είμαι αντίθετο στο να ανακαλέσω αυτές τις τροπολογίες που έχω καταθέσει, να βάλουμε όμως την ιδέα της δημιουργίας μιας ομάδας μελέτης, η οποία θα ασχοληθεί με αυτό το στόχο. Για την επόμενη τριετή αναθεώρηση του καονισμού δηλαδή. Αφού δούμε τις δυσκολίες, ε, με τις αντιθέσεις που υπάρχουν κτλ. Να δημιουργήσουμε λοιπόν μια ομάδα εργασίας που θα μελετήσει το στόχο χορήγησης απαλλαγής με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Δεύτερη, ο δεύτερος λόγος που παίρνω τον λόγο. Ε, στην ε, Επιτροπή Βιομηχανίας συζήτησα με άλλου ευρωβουλευτές και θα ήθελα να λάβετε υπόψη σας στους συμβιβασμού τις ε, τροπολογίες της Επιτροπής Βιομηχανίας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλφιν. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Όχι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα απλώς εν συντομία να σχολιάσω δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα θέλω να συμπορευθώ με όλους τους άλλους οι οποίοι ευχαρίστησαν τον εισηγητή για τα νέα έγγραφα εργασίας που μας έχουν δώσει και ένα έγγραφο που περιλαμβάνει τις πιο συχνά ερωτώμενες ερωτήσεις. Θα ήθελα τώρα να κάνω και ένα σχόλιο. αντί να έχουμε μονάχα εφαρμοστικές πράξεις, θα έχουμε και κατεξουσιοδότηση πράξης. Θέλω να σας πω ότι όλες αυτές οι διαδικαστικές κατεξουσιοδότηση πράξης περιλαμβάνουν και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντίθετα με τις προηγούμενες. Επομένως, αυτά τα οποία παραμένουν για να αποφασιστούν από την Κομισιόν μπορούν να τύχουν απόφαση μόνο εάν υπάρχει σιωπηρή έγκριση του Κοινοβουλίου και εάν το Κοινοβούλιο θέλει να κάνει κάποια άλλη τροποποίηση, αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή, η ίδια η χρήση των κατεξουσιοδότησης πράξεων για το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτό το στοιχείο γιατί οι εφαρμοστικές πράξεις δεν είναι πια υπόθεση μόνο της Κομισιόν χωρίς την έγκριση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Και επίσης αναφερθήκατε στη διαδικασία λέγοντας ότι είναι μια επαχθής διαδικασία. Δεν είναι και τόσο επαχθής στο κάτω-κάτω της γραφής. Έχετε δύο δυνατότητες. Μία η οποία απαιτεί μια διαδικασία τριών εβδομάδων που υπάρχει ο χρόνος αντίδρασης από το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι με τις πράξεις εξιοδότησης έχουμε κάτι το οποίο αυξάνει σημαντικά τις δυσκολίες λήψεως αποφάσεων. Ένα δεύτερο θέμα που θέλω να αναφέρω έχει να κάνει με τα άθρα τα οποία συνδέονται με τα χρηματοδοτικά μέσα. Και, στο, και πάλι στο έγγραφο αυτό που έχετε παρουσιάσει σε σχέση με τις συχνές ερωτήσεις αναφερόσαστε στην ανάγκη να υπάρξει μια εξάντε πληροφόρηση του Κοινοβουλίου σε σχέση με τους κινδύνους χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα παραπάνω που θα πρέπει να μας υποχρεώσει να σκεφτούμε καλύτερα τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί το Κοινοβούλιο μπορεί να πληροφορηθεί, αλλά τι θα γίνει όταν πληροφορηθεί. Το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να είναι το θεσμικό όργανο το οποίο αποφασίζει σε σχέση με την εκτίμηση κινδύνου. Ακόμα και αν πληροφορούμαστε για κάτι, τι θα προκύψει στη συνέχεια. Ένα ακόμα παράδειγμα λοιπόν που το Κοινοβούλιο χρειάζεται πληροφορίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε δράση από τη μεριά του Κοινοβουλίου και όχι απλώς μια εξάντε πληροφόρηση. Για την ε, ανάλυση της πληροφορίας εκ των υστέρων, εξ δηλαδή και όλα αυτά, σίγουρα πρέπει να έχουμε μια πλήρη πληροφόρηση. Αλλά εξάντε απλώς να έχουμε κάποιες πληροφορίες οι οποίες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αντιδράσουμε αν αυτό είναι απαραίτητο για τη χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων. Είναι λοιπόν ένα παράδειγμα. Έχω και άλλα παραδείγματα σε σχέση με τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι θα θέλανε να λάβουν το λόγο σε αυτό το στάδιο. Στρέφομαι λοιπόν προς την Επιτροπή, εάν θέλει να λάβει το λόγο. Κύριος Σταβένα, κύριος Παραντή, δεν θέλετε να κάνετε παρατηρήσεις. Κύριος Παραντή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί από τους διάφορους κοινοβουλευτικούς, τους αξιότιμους κύριους κοινοβουλευτικούς. Και αναφέρομαι και στην κυρία Γκρέσλε, το, το βασικό θέμα που ετέθη αφορούσε τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Είναι τρόποι εφαρμοστικοί, δηλαδή είναι διαδικασίες εφαρμογής. Θα πρέπει να ακολουθηθεί μια νέα διαδικασία, η οποία είναι αυτή η οποία προβλέπεται στη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνήθως αυτό σημαίνει μια απόφαση της Κομισιόν μετά από ενισχυμένη συνεργασία και διαβούλευση με το Συμβούλιο αλλά και το Κοινοβούλιο. Εγώ διαπιστώνω ότι πράγματι αυτά τα οποία θα μεταφερθούν από τις τωρινέ διαδικασίες εκτελεστικού χαρακτήρα στο νέο δημοσιονομικό κανονισμό είναι μια μικρή δέσμη ρητρών και έχουμε εργαστεί πάρα πολύ με την κυρία Γκρέσλε για τα θέματα αυτά και έχουμε προτείνει στην εισηγήτρια μια σειρά από διατάξεις στις, στον τωρινό δημοσιονομικό κανονισμό που θα πρέπει να μεταφερθούν <clears throat> στο νέο κανονισμό. Υπάρχουν κάποια άρθρα για τα οποία πρέπει να υπάρξει ακόμα συζήτηση. Συμφωνούμε μαζί της, συμφωνούμε για να μειώσουμε αυτά τα οποία θα περιλαμβάνονται στο δημοσιονομικό κανονισμό και όχι στις εφαρμοστικές διατάξεις. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε τους ίδιους στόχους να θέσουμε στο δημοσιονομικό κανονισμό μόνο τα ουσιώδη και να αφήσουμε στις κατεξουσιοδότης πράξεις μόνο αυτά τα οποία αποτελούν ένα συμπλήρωμα, μια διευκρίνηση, μια σειρά από σε σχέση με το θέμα το οποίο καλύπτει η κάθε πράξη. Για να απαντήσω δε στον κύριο Μιλντερ, αυτά που είπε για το γιατί είναι τόσο δύσκολο να αλλάξουμε το δημοσιονομικό κανονισμό. Όχι κύριε Μιόλτερ, δεν είναι δύσκολο, είναι μια νομοθετική πράξη, ακολουθεί λοιπόν τη διαδικασία που λέγαμε τα παλιά τα χρόνια συναπόφασης. Είναι κάτι το οποίο είναι ίσως πιο βαριά διαδικασία από μια τροποποίηση των εφαρμοστικών πράξεων, δηλαδή της, των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση. Αλλά επειδή η διαδικασία συναπόφασης μπορεί να ακολουθήσει πολλούς δρόμους, πρώτη ανάγνωση, δεύτερη ανάγνωση, ακόμα και τρίτη ανάγνωση, είναι σαφές ότι μπορεί να υπάρξει μια τροποποίηση, αλλά αυτό απαιτεί κάποια χρονική διάρκεια και ίσως δεν είναι το πιο πρόσφορο, πιο πρόσφορος τρόπος εάν είναι νέε οι συνθήκες οι οποίες προκύπτουν και χρειάζεται μια ταχεία αλλαγή. Γι' αυτό προτείνουμε στην κυρία Γκρέσλε να προσπαθήσει να κρατήσει ε, στις εφαρμοστικές πράξεις τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη ευελιξία. Και εδώ αναφέρομαι στα κατόφλια. Υπάρχουν πολλά κατόφλια τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν ε, επί τη βάση των οικονομικών συνθήκων και συγκυριών. Παραδείγματο χάρη, τα κατόφλια για τις διαδικασίες που αφορούν τα ακίνητα που προτείνονται, από, που προτείνονται τώρα από την εισηγήτρια μαζί με την κυρία Όλ Μάιερ. Υπάρχουν δύο κατόφλια 200.000 και 5 εκατομμύρια, αλλά αυτά μέσα στο χρόνο μπορούν να τροποποιηθούν σαν συνάρτηση της ε, εξέλιξης των τιμών των ε, ακινήτων και επομένως θα πρέπει να μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτά τα κατόφλια με ένα πιο γρήγορο τρόπο. Αυτό το οποίο μας ε, δυσκολεύει στις κατεξουσιοδότηση πράξεις είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να απασχολήσει και το Κοινοβούλιο. Για μας υπάρχει μια σειρά από διατάξεις που προβλέπονται από την πρόταση των εισηγητών που κατά την άποψή μας αντιφάσκουν προς τη συνθήκη και προς το δικαίωμα πρωτοβουλίας, το αποκλειστικό δικαίωμα πρωτοβουλίας της Κομισιόν. Πρέπει να δούμε τις τροπολογίες 210, 214, 219 καθώς και άλλες, οι οποίες προσπαθούν να επιβάλλουν μια διαδικασία σχεδόν νομοθετικού χαρακτήρα για τις κατεξουσιοδότηση πράξης και αυτό φυσικά αντιβαίνει με την ε, Συμφωνία Κοινή Κατανόησης όπως λέγεται, η οποία υπεγράφει και από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου μαζί με τον πρόεδρο της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Πιστεύω λοιπόν ότι η τροπολογία 213 αντιβαίνει απόλυτα στο πνεύμα αυτής της συμφωνίας. Αυτό το οποίο επιζητούμε εμείς από την δική μας πλευρά είναι να ακολουθήσουμε το άρθρο 290 και την κοινή κατανόηση και να μην ακολουθήσουμε μία κατεύθυνση η οποία θα αντιβαίνει στην συμφωνία αυτή κοινή κατανόησης. Είναι προφανέ, βέβαια ότι η συνεργασία που έχουμε με του εισηγητέ και με του άλλου βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θέλουν να συμβάλλουν στην εκπόνηση αυτού του νομοθετήματο για την εξουσιοδότηση πράξη. φυσικά θα παραμείνει πολύ στενή συνεργασία. Αλλά θέλουμε να διατηρήσουμε <clears throat> το κείμενο τη κοινή κατανόηση και τι διατάξει τη συνθήκη για την ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην παραβιαστεί το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Κομισιόν. Αυτά για τις κατεξουσιοδότησες πράξεις. Και το άρθρο 56 η κυρία Γκρέσλερ είπε ότι υπήρχαν πολλές προτάσεις για το άρθρο 56, πολλές τροπολογίες. Εγώ ήμουνα παρόν στην Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η συμβαστική λύση που φαίνεται να επικρατεί και ίσως θα ψηφιστεί σήμερα το απόγευμα είναι σε γενικέ γραμμέ αποδεκτή, αποδεκτή από την Κομισιόν και μπορεί αυτή να αποτελέσει και μια θέση διαπραγμάτευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εναντί των κρατών μελών που, των κρατών μελών που δεν συμφωνούν ιδιαίτερα με την πρόταση της Κομισιόν για τα θέματα αυτά και δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Υπάρχει κάτι ακόμα το οποίο θέλω να πω σε σχέση με αυτή την πρόταση που αρχίζει να αναδύεται. Το θέμα της ε, διαπίστευσης της Κομισιόν μέσα στα συστήματα ελέγχου των κρατών μελών υπάρχει το θέμα της ε, διχοτομίας μεταξύ του Σαλ και ΜΕΙ στα αγγλικά. Λένε ορισμένα κείμενα ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ε, αξιολογήσει τα συστήματα ελέγχου στα κάθε μελη Μία τέτοια διατύπωση μας φαίνεται ότι είναι αντιπαραγωγική. Αν η Κομισιόν θέλει να αξιολογήσει αυτά τα συστήματα επειδή το ζητά ένα κράτος μέλος, το κράτος μέλος θα μπορούσε να μην επιζητήσει να έχει ένα σωστό σύστημα γιατί θα έλεγε ότι με τον τρόπο αυτό η Κομισιόν θα το διορθώσει και να πετάξει τον μπαλάκι στην Κομισιόν η πείρα μας από τον προγραμματισμό μέχρι στιγμής δείχνει ότι αν, εμεί πρέπει να επαναξιολογούμε συστηματικά όλα τα συστήματα ελέγχου πρωτού αρχίσουν να λειτουργούν στα κράτη-μέλη, θα υπήρχε κίνδυνος μεγάλης καθυστέρησης για τα διαφορετικά ταμεία. Επομένως για μας θα πρέπει να είναι η διατύπωση The Commission may appraise. Μπορεί να αξιολογήσει τα συστήματα και βλέπω ότι και η κυρία Γκρέσλα στην τροπολογία 313 συμφωνεί με την διατύπωση αυτή. Αυτά για το άρθρο 56. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά ήταν τα σημεία για τα οποία ήθελα να απαντήσω. Εάν μου επιτρέπετε τώρα, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο, να κάνω μερικές γενικές παρατηρήσεις. Ε, θέλω να έρθω σε μερικά σημεία τα οποία είπαν ορισμένοι κοινοβουλευτικοί. Εμείς <clears throat> θεωρούμε ότι σε ορισμένε περιπτώσεις ο, οι εισηγητές παραπέμπουν σε νομικές βάσεις, σε πράξεις τομεακού χαρακτήρα, μια σειρά από δεσμεύσεις οι οποίες θα εφαρμοζόντουσαν στην Κομισιόν σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Για παράδειγμα, υπάρχει τροπολογία 68 για το άρθρο 55 που αφορά τους ε, εντολοδόχους, δηλαδή τους φορείς τους οποίους η Κομισιόν μπορεί, τους οποίους μπορεί να εξουσιοδοτήσει για την εκτέλεση ενός τμήματος του προϋπολογισμού. Στο άρθρο αυτό 5.5 και το έχει και στον πίνακα της η κυρία Γκρέσλε που θα τον κοιτάξω προσεκτικά τώρα, λέγεται ότι η Κομισιόν θα πρέπει και τον προτέρων να έχει καθορίσει ποιο είναι ο στόχο ο οποίο επιζητείται, ποια είναι τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, ποιε είναι οι μέθοδοι εκτέλεση και πολλά άλλα τα οποία θα πρέπει να καθορίζονται από την βασική πράξη χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος του περίοδου προγραμματισμού. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα βαριά σαν διαδικασία και <clears throat> υπάρχουν πράξεις χρηματοδότησης που έρχονται σε γνώση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που δίνουν τις ίδιες πληροφορίες αλλά όχι στο βασικό νομοθετικό κείμενο αλλά είναι μέσα στα πλαίσια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οι εισηγητές επανέρχονται σε αυτή την πρόταση, στην τροπολογία 306. Αλλά προστίθενται στις, ε, στην υποχρέωση της Κομισιόν να έχει αυτά τα στοιχεία ήδη στη βασική πράξη. Γι' αυτό έχουμε πρόβλημα με την τροπολογία 68, γιατί προβλέπει πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνονται καταρχήν στη βασική πράξη. Το ίδιο για την ε, τροπολογία 67 που αφορά το άρθρο 130 για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και μας ζητείτε να προβλέψουμε πάρα πολλά πράγματα εκ των προτέρων και θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να μας εμποδίσει να έχουμε μια σωστή προσαρμογή σε ρευστές ε, συνθήκες, ιδίως όταν μιλάμε για μια τόσο μακρά περίοδο προγραμματισμού, 7 χρόνια. Η τροπολογία 424 επίσης ε, έρει ορισμένες διατάξεις και κάνει πιο άκαμπτη τη διαδικασία του προπολογισμού και ακόμα ένα κούτσικο λεπτό θα ήθελα να λάβω το λόγο σε σχέση με κάποιες τροπολογίες που αφορούν τις μεταφορές πιστώσεων. Τροπολογία 22 για το άρθρο 23 κυρίως και πάλι η Κομισιόν αυτό το οποίο θέλησε να επιτύχει είναι μια κάποια ευκαμψία για τη διαχείριση των διοικητικών πιστώσεων μεταξύ των γενικών διευθύνσεων. Δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα μετακίνηση των κονδυλίων Πριν από 10 χρόνια, πριν να περάσουμε στον προπολογισμό από τη βάση δραστηριοτήτων, υπήρχε ένα διοικητικό προπολογισμό, ο οποίο μπορούσε να αντιμετωπιστεί όπω ήθελε να το κάνει η Κομισιόν και επί τη βάση των διοικητικών αναγκών. Τώρα είναι ε, διηρημένος σε διάφορους επιμέρους προπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων για να μπορούν να κατανέμονται τα κονδύλια στι διάφορε γενικέ διευθύνσει. Υπάρχουν θετικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτό, αλλά θα θέλαμε και κάτι περισσότερο. Μια άλλη πτυχή, η οποία είναι πολύ σημαντική, είναι αυτή των πιστώσεων πληρωμών και εκεί πάλι για τι πιστώσει πληρωμών. Στον βαθμό που πρόκειται για πιστώσει που θέλουμε να, τις, να τα κατευθύνουμε τα ποσά αυτά εκεί που είναι η καλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων, αν υπάρχει ένας τομέα, όπου μπορούμε με μετακίνηση κονδυλίων να επιταχύνουμε την εκτέλεση του προϋπολογισμού και εκεί αυτή η άποψη δεν έχει γίνει δεκτή από, τους από την εισηγήτρια με ένα επαρκή τρόπο και επομένως υπάρχει τροπολογία 266 η οποία παρόλα αυτά θα επέτρεπε να γίνεται αυτή η πιο εύκολη μεταφορά κονδυλίων εάν οι αρχές του προϋπολογισμού δεν προέβαλαν ένσταση μέσα σε τρεις εβδομάδε. Μία ακόμα παρατήρηση, επειδή η κυρία Όλ και Μάιερ είναι παρούσα για τα θέματα των ακινήτων. Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος κοινοβουλευτικός σε αυτές τις διαδικασίες για τα κίνητα που υπάρχει εξάλλου στον ισχύοντα κανονισμό. Διαπιστώνουμε φυσικά με μεγάλη ικανοποίηση ότι το Κοινοβούλιο ε, ικανοποίηση χωρί έκπληξη ε, ότι το Κοινοβούλιο συμφωνεί με μας ε, να χρηματοδοτούμε τα κινητά με δάνεια. Αλλά το να πρέπει να ερχόμαστε στην Επιτροπή Προπολογισμού, ε, στην Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών σε τρει διαφορετικέ φάσει, πριν το διαγωνισμό, πριν να υπογράψουμε τη σύμβαση, νομίζω ότι αυτό μάλιστα θα έβλαπτε και τη σύναψη της σύμβασης με τον ανάδοχο. Όλα αυτά θα δημιουργούσε μια επαχθή διαδικασία. Αν μπορούσαμε λοιπόν κάποια στιγμή να βρούμε μια διαφορετική τροπολογία, να υπάρχει μια εξέλιξη αυτή την τροπολογία. Κάτι άλλο που μας φαίνεται σημαντικό. Αν η πρόταση της Κομισιόν που αφορά την ενοικίαση ακινήτων ε, ε, οδηγήσει στην μείωση του ενοικίου, μειώσει λοιπόν τα έξοδα, τότε φαντάζομαι ότι η Δημοσιονομική Αρχή δεν θα έχει ανάγκη να γνωρίζει πριν το διαγωνισμό, πριν από την ε, σύμβαση, τι θα προτείνουμε. Γιατί δεν θα υπάρχει αύξηση των δαπανών. Και θα τελειώσω με το εξής. Όντως, σε ορισμένε περιπτώσεις ε, έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχουν αιτήματα για reporting, για σύνταξη αναφορών υπερβολικά. Παραδείγματο χάρη, ε, τροπολογία 48 ε, για το άρθρο 34. Πρέπει να κάνουμε μια έκθεση για, την, ε, για τον κατάλογο των ε, επιχειρήσεων που εκτελούνται από όλους τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 55 οι κοινοτικοί οργανισμοί του άρθρου 185, οι agencies, ε, οι οργανισμοί δηλαδή, οι, οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, ήδη στην έκθεσή μας για αυτές τις απλές, ε, για αυτούς τους ε, οργανισμούς, η έκθεσή μας είναι 500 σελίδες. Αν προσθέσουμε ακόμα τον κατάλογο όλων των επιχειρήσεων, των υπολείπων ε, που, εκτελούν κάποια έργα κατανάθεση από την Κομισιόν, θα ξεπεράσουμε, την έκθεση, θα, θα ξεπεράσουμε τις χίλιες σελίδες στην έκθεση. Δεν νομίζω, δεδομένη στις πίεσεις χρόνου που έχετε, ότι θα μπορείτε να διαβάζετε τις εκθέσεις. Και εσείς και η Επιτροπή Προπολογισμών. Αυτά. Ε, σας ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα και σας ευχαριστώ που μου αφήσατε τον λόγο τόση ώρα. Θα είμαι πολύ πιο σύντομος από τον Ερικ Παραντή. Έχω λιγότερα πράγματα να πω για τη διαδικασία απαλλαγή. Χαιρετίζω την τιμιότητα και το θάρρος του κυρίου Ντί και θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καταλαβαίνω το πολιτικό νόημα του να υπάρχει ε, μία απαλλαγή την επόμενη χρονιά, μετά τη χρονιά δηλαδή της εκτέλεσης. Αλλά η απαλλαγή βασίζεται ε, στην έκθεση του συνεδρίου. Θα μπορούσαμε να έχουμε του λογαριασμού λίγο πιο πριν. Αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε μια μέθοδο εργασία με το ελεκτικό συνέδριο, ούτω ώστε να ελέγχονται οι λογαριασμοί πιο γρήγορα, αλλά ακόμα πιο σημαντικό, το βασικό στοιχείο για ένα πιο σύντομο χρονοδιάγραμμα θα ήταν ε, ο έλεγχο των συναλλαγών. Για να μπορέσει το ελεκτικό συνέδριο να δώσει μια γνωμοδότηση υψηλή ποιότητα, θα πρέπει κατά ανάγκη να κάνει μια δειγματοληψία κατά τη διαδικασία της χρονιάς εκτέλεσης. Αν τώρα θα έπρεπε η, το χρονοδιάγραμμα αυτό να συμπιεστεί, τότε θα ήταν αναγκασμένο το ελεκτικό συνέδριο να κάνει πιο νωρίς τη δειγματοληψία. Αυτό θα, ήταν, θα σημαίνει ότι θα είναι πιο λιγότερο αντιπροσωπευτικό και επομένω η ποιότητα του ελέγχου θα ήταν χειρότερη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτά τα πράγματα έτσι εντάχει. Νομίζω ότι η επιλογή του κυρίου Ντί είναι πολύ λογική, αλλά θα πρέπει τα θεσμικά όργανα, κυρίως η Κομισιόν και το Ελεγκτικό Συνέδριο, να βρουν μια άλλη μέθοδο εργασίας, η οποία θα μπορέσει να εξασφαλίσει την ε, επιβράχηση της διαδικασίας. Τώρα, για το θαυμάσιο χρωματιστό πίνακα της κυρίας Γκρέσλε. θέλω να πω ότι Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακή, εντυπωσιακός αυτός ο πίνακας, αλλά διαρωτώ με τι στην οργή είναι αυτή η ιστορία. Σε ό,τι αφορά α, τους τρόπους εκτέλεσης, αυτή είναι το, μια ανθιπολεπτομέρεια. Το υπόλοιπο είναι οι κανονισμοί, οι τομεακοί. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι αυτό που έχει σημασία πάνω απ' όλα είναι ότι δεν έχουμε όλοι τις ίδιες προτεραιότητες με την Επιτροπή προπολογισμού και την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ε, ευχαριστώ κύριε Ταβέρν και κύριε Παγαντή. Α, νομίζω ότι τώρα την ε, προκαλέσατε την κυρία Ντεμαγιέρ και θέλει να απαντήσει. Όχι. Ε, δεν είναι καλό να με τσιγκλίσετε γιατί και εγώ θα αντιδράσω. Τώρα, επί της ουσίας, καταρχήν η κτηριακή πολιτική, η πολιτική ακινήτων της Κομισιόν μέχρι πριν από 2-3 χρόνια ε, δεν ήταν και η διαφανέστερη. Δεν ε, γινόταν να είναι διαφανής έτσι όπως ήταν. Στις πρώτες συζητήσεις με την Κομισιόν, μία καθήλυνα αρμόδια της Κομισιόν μας είπε την άποψη ότι τα κτίρια στο βαθμό που κινούνται στα πλαίσια των τίτλων του προϋπολογισμού, κάπως έτσι το διατύπωσαν, δεν θα έπρεπε να αλλάξουν θέση. Μετά ρώτησα ένα κτίριο 600 εκατομμυρίων αν είναι στα πλαίσια του τίτλου τι θα έπρεπε, πώς θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί και είπε αν μπορεί να ε, γίνει ε, στα πλαίσια του προϋπολογισμού θα βάλουμε τα 600 εκατομμύρια εκεί και μετά ζήτησα τον, τον ε, κατάλογο των κτηρίων που μπορούσαν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά και είχε 40 εκατομμυρίων αξία κτίρια εκεί, δηλαδή με μεγάλη επίδραση στον προπολογισμό. Άρα θα πρέπει να έχουμε σαφείς ορισμούς, να επιμείνει το Κοινοβούλιο εκεί. Τώρα, για τις τρεις τροπολογίες. Ε, αν ζητήσω σε τρία σημεία πληροφορίες, δεν σημαίνει ότι τρεις φορές θα ζητήσω από εκεί την ε, άδεια. Πρέπει να υπάρχει κοινοποίηση αν δεν μπορεί πια να αποφασίζει τίποτε το Κοινοβούλιο. Αν έχουν δηλαδή, όταν έχουν τελειώσει τα πάντα, τρίζοντας τα δόντια, ε, λέει το Κοινοβούλιο, α, δόθηκαν τόσα εκατομμύρια που και εμείς δεν μπορούμε ούτε να γνωμοδοτήσουμε. Γι' αυτό η γνώμη μου και η γνώμη των άλλων με τους οποίους διαβουλεύτηκα είναι να γίνεται μια σύντομη ενημέρωση για τα προγραμματιζόμενα έργα, να τα συζητήσουμε ως Κοινοβούλιο, ούτως ώστε να μπορούμε να λέμε τη γνώμη μας, είτε θετική ή επικριτική ή όποια θέση τέλος πάντων, δεν θα είναι μια τεράστια διαδικασία, τελείως απλή, αντιγραφειοκρατική. Εκείνο που είναι σημαντικό θεωρώ είναι τα στοιχεία τα οποία θα συμπεριλαμβάνει η κοινοποίηση θα είναι αξιόπιστα και όχι εκ των υστέρων να διαφέρουν ε, κατά εκατομμύρια και εκ των υστέρων να δηλώνονται αν δηλωθούν, γιατί τότε δεν θα χρειάζεται πια καμία ε, κοινοποίηση. Απλώς θα πρόκειται για μια καθαρά πράξη ε, εντελώ μη δεσμευτική. Επίσης, η Κομισιόν αναφέρει ρητά την μικροδιαχείριση, ότι θα την επηρεάζαμε. Όχι, δεν το κάνουμε αυτό, για να μην πω ότι εμείς είμαστε ένας ε, φορέας exposed. Εγώ, ως ε, μέλος του, της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμών, θέλω να μην είμαι εκ των υστέρων ε, μια, ένας φορέας παρακολουθήσεις και ελέγχου. Θέλω να ξέρω τι γίνεται. Αν πηγαίνουν κάποια κονδυτικό που μπαίνουν εκεί λόγω κάποιων παρατηρητιών στα θέματα των κτηρίων, τι νόημα έχει να κάνω έλεγχο εκ των υστέρων. Πρέπει εκ των προτέρων να ξέρω τις προϋποθέσεις και τη λειτουργία και να ε, γνωμοδοτήσω. Πράγμα που προβλέπεται και στο δημοσιονομικό κανονισμό. Δεν μπορεί εκ των υστέρων όταν έχουν συναυθεί συμφωνίες 30 χρόνων ε, αφού συναυθεί η συμφωνία να την ε, κριτικάρω, διότι στα δύο χρόνια, διότι ακόμα θα συνεχιστεί 28 χρόνια και εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα στη σύμβαση αυτή. Οπότε δεν έχει καθόλου νόημα. Επίσης, ε, κρυφογελώντας, ε, σημείωσα ότι είπατε ότι με ε, ικανοποίηση παρακολουθούμε σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις του Κοινοβούλιο είχε πει στον τομέα των κτίριων να διευκολύνονται τα δάνεια διότι η αδιαφάνεια και η συνθετότητα των κερδών των ενδιάμεσων θα πρέπει να τερματιστεί κάποια στιγμή. Είχαμε πολλά τέτοια περιστατικά. Δεν θα παραθέσω κάποια από αυτά. Πάντως θέλουμε σαφή και ξεκάθαρη και διαφανή χρηματοδότηση των κτίριων. Λέει μετά πρέπει να διαγράψουμε στο εδάφιο αυτό μια πρόταση στην οποία προβλέπουμε ένα ενδεδειγμένο χρονικό διάστημα της ε, ε, ε, ολοκληρωτικής ε, χρηματοδότησης της, όλης της καταβολής. Ε, Έψαξα να βρω αν υπάρχει αυτό. Το βρήκα σε 10 κρατημέλη. Το ενδεδειγμένο χρονικό διάστημα μπορώ να πω και σταθερό. Δεν ξέρω. Εκείνο που θέλουμε να πούμε είναι ότι όταν κάποιος ε, παίρνει ένα δάνειο θα πρέπει να είναι σαφές πότε θα αποπληρώσει. Δεν θέλουμε η Κομισιόν να γράψει ότι, ε, να, να μας πει ότι αυτό το κομμάτι για την αποπληρωμή θέλουμε να το βγάλουμε και ότι τα δάνεια θα πρέπει να διατηρούνται ε, για κάποιο χρονικό διάστημα προσδιορίστο. Θέλουμε σαφείς ε, προδιαγραφές σε σχέση με την ε, κτηριακή πολιτική και την αποπληρωμή των δανείων. Και το τρίτο βήμα, πολύ σημαντικό, διότι εγώ ε, ως εισηγήτρια έχω μια διετή εμπειρία και έχω να παρατηρήσω το εξής διαπίστωσα ότι οι ε, κοινοποιήσει γίνονται εφόσον εγώ στον μετέπειτα έλεγχο διαπίστωσα ότι δαπανήθηκαν πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι αυτά που μας είχαν αρχικά να κοινοποιηθεί. Οπότε το τρίτο βήμα σημαίνει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να υποβάλει και μια έκθεση που θα λέει τι ακριβώς στήχησε το κτίριο και ποιες είναι, ποιες ήταν οι οριστικές, οι οριστικοί όροι για τη χρηματοδότηση. Και μετά αυτό θα είναι το τρίτο βήμα μετά από την ε, ε, σχετική σύμβαση. Αυτό μπορεί να μας το δώσουν ενημερωτικά. Δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Επίσης υπάρχουν τέτοιες, τέτοιοι εθνικοί κανόνες σε αρκετά κράτη-μέλη. Η Κομισιόν ε, θα πρέπει να παρακολουθεί το θέμα πολύ περισσότερο, δηλαδή απαιτούνται πολλά περισσότερα από την Κομισιόν από ότι το Κοινοβούλιο, γιατί θα πρέπει να έχει μια διαφανή πολιτική ακινήτων, που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο όμως να γίνει αυτό το πράγμα. Και έχω λάβει υπόψη μου τις παρακλήσεις των συναδέλφων πολύ σοβαρά που επανειλημμένα, διαπαραταξιακά μου έχουν παραπονεθεί ότι η πολιτική για τα ακίνητα ε, ε μας κοινοποιείται καθυστερημένα με αδιαφανή τρόπο πολλέ φορέ και χωρίς να ανταποκρίνεται στην τάξη, στο, στο μέγεθος του κτηρίου. Δισεκατομμύρια ε, μπορεί να χάνονται ε, σε σχέση με την κτηριακή πολιτική. Οπότε χρειάζεται μια διαφάνεια και καλύτερη οργάνωση. Ευχαριστώ κύριε Αλμάιερ. Θα δώσω σύντομα το λόγο στους δύο συγκητές αν το επιθυμούν για να απαντήσουν. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι Υπάρχουν διάφοροι που θέλουν να φύγουν, γιατί θα γίνει σοφορία στην, Επιτροπή, Περιφερειακή Επιτροπή. Επομένω, οι δύο εισηγητέ ε, μπορούν να δώσουν μια σύντομη απάντηση, αλλά θα, θα τα ξαναπούμε στι 13. Δεν τελειώνει τώρα η συζήτηση. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Κυρία Ολμάρια. το παρουσίασε πάρα πολύ σωστά το θέμα αυτό. Είτε είμαστε η κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ευρώπη, είτε όχι. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι εδώ πρόκειται για μια περί περίπτωση ε, εισαγωγής της συναπόφασης για τα θέματα αυτό, αυτό το οποίο έγινε με την ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Είπε τώρα ή ποτέ ο κύριος Μίλτερ, γιατί πράγματι τώρα είναι η στιγμή που μπορούμε πράγματι να εφαρμόσουμε το άρθρο 290. Υπάρχουν ουσιαστικές διατάξεις. Οι ουσιαστικές διατάξεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο νομικό κείμενο αυτό καθε αυτό. Η στιγμη που μπορουμε πραγματι να εφαρμοσουμε το αρθρο 290 υπαρχουν ουσιαστικες διαταξεις οι ουσιαστικες διαταξεις θα πρεπει να περιλαμβανονται στο νομικο κειμενο αυτο καθεαυτό. η κομισιον έχει αναφέρει 12 τέτοιες ουσιώδεις ρήτρες, εμείς έχουμε βρει άλλες 8 και το σύνολο επομένω των ουσιωδών στοιχείων είναι 20. Η Κομισιόν θέλει επομένω ε, κάτι περισσότερο να τονίσει σε αυτό το θέμα από ότι εμείς. Εμείς είχαμε 8 τέτοιες προτάσεις, η Κομισιόν 12. Εγώ όμως δεν ξέρω τι από όλα αυτά θα πρέπει να τεθεί σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Κάρφιν είναι σημαντικό. Πώς θα ρυθμίσουμε τα θέματα των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ή τις δεχόμαστε ή δεν τις δεχόμαστε καθόλου. Εμείς αυτό το οποίο προτείνουμε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη σύγκρουση. Αν δεν υπάρχει λοιπόν κάποια διαφορά απόψεων, μπορούμε να έχουμε εύκαπτους κανόνες. Τι γίνεται όμως όταν υπάρχει κάποια διαφωνία. Θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε και να αλλάξουμε τους κανόνες και να τους ξαναφτιάξουμε από την αρχή ή θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Εμείς προτείναμε έναν δρόμο τον οποίο η Κομισιόν αυτή τη στιγμή τον απορρίπτει. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι εγώ έχω δεχτεί την πιο ε, αδύναμη νομική θέση. Μια θέση που δεν μας επιτρέπει να απορρίψουμε ούτε να δεχτούμε πλήρως αυτές τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξη. Είναι λοιπόν κάπως αποδυναμωμένη η νομική μας θέση για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Γι' αυτό εγώ είχα ζητήσει να είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε τις προτάσεις της Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Νομίζω θα ήταν σωστό λοιπόν στην περίπτωση να σκεφτούμε περισσότερο για τα χρηματοδοτικά μέτρα μέσα. Έχουμε πολλές φορές συζητήσει για τα θέματα του κινδύνου και της αστικής ευθύνης στον προϋπολογισμό. Όταν κάθε χρόνο ένα 10 με 15% του προϋπολογισμού περνάει από τα χρηματοδοτικά μέσα και μόνο 3% αντιμετωπίζει προβλήματα, αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα λειτουργούν σε κάποιο βαθμό. Αλλά το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε στις εκλογές μας ότι εμείς προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε τους ε, κίνδυνους. Νομίζω ότι ήταν απόλυτα λοιπόν εξισορροπημένο και μετριοπαθές αυτό το οποίο θέλησαμε εμείς να κάνουμε. Έχουμε τώρα τις γνωμοδοτήσεις της Ήτρε, της ΑΦΕΤ ε, και της ε, Ρέγγι της Επιτροπής ε, Περιφερειακών Θεμάτων. Ίσως θα πρέπει να δώσουμε κάποιο βραβείο ομορφιά σε ορισμένες τροπολογίες που έχουν κατευθεί από αυτές τις νομοθετικές επιτροπές. Γιατί εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω πολύ καλά τι ζητούν αυτές οι, οι τροπολογίες. Αν η Κομισιόν θέλει να ελέγχει αυτή πλήρως τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Ταμείου, αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί πράγματι να το εννοεί ότι αυτό θέλει. Αν έχουμε κάνει εμεί τόσο άσχημα την εργασία μας που να έχουμε χάσει βασικά στοιχεία, ναι. Αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι βασικοί δημοσιονομικοί κανόνες και τους οποίους θα πρέπει να τηρήσουμε. Θα πρέπει να ζητήσω λοιπόν από όλους τους συναδέλφους γιατί ε, θα πρέπει να σκεφτούμε και ορισμένε από τι τροπολογίε τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που, κατά τη δική μου άποψη, είναι και επικίνδυνε για όλο το δημοσιονομικό οικοδόμημα και θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτέ. Ευχαριστώ. Ο κ. Ριβελίνη, τα τελευταία λόγια. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Μετά από την κυρία Γκρέσλερ, ε, θέλω να, κάνω ένα προσωπικό σχόλιο. Όταν είμαστε ε, στην αίθουσα συνεδρίασης και, ακούμε όλους τους ενδιαφερόμενους για το θέμα. Όλοι, όλοι θέλουμε και το λέμε να μειωθεί η γραφειοκρατία, να υπάρξει μεγαλύτερη ενάργεια ε, και με καλύτερος και πιο ποιοτικό έλεγχος. Αλλά όταν μαζί με την Γκρέσλερ ε, είμαστε εδώ σε αυτή την αίθουσα, όλες αυτές οι προθέσεις που όλοι τις ε, συμμερίζονται σε αυτή την ε, αίθουσα ξαφνικά αλλάζουν. Λες και έχουν μια άλλη βούληση, όχι αυτή που εκφράζουν. Ε, εμείς τα, είπαμε τον κύριο Οντί. Καταρχάς έχουμε μια ιστορική ευκαιρία για δύο λόγους. Καταρχάς η συνθήκη της ε, Λισαβόνας και δεύτερον γιατί έχουμε στο πλευρό μας την ικανότατη κυρία Γκρέσλερ που ε, συνεισφέρει τα μάλα για να, και κάνει ό,τι μπορεί για να πλουστεύσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και για να βελτιώσουμε τον έλεγχο. Το τελευταίο. Ο σεβασμός του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει πάντα να το προτάσουμε αυτό το θέμα. Να υπάρχει σεβασμός και από το Συμβούλιο και από την Κομισιόν, γιατί είναι κεντρικό όργανο. Όπως είπε η κυρία Γκρέσλερ, η δουλειά μας ούτως ή άλλως ελέγχεται οποιοδήποτε έρχεται εδώ στο Κοινοβούλιο μπορεί να μας ελέγξει. Και μπορεί να μας ελέγξει οποιοδήποτε άνθρωπος εκπροσωπείται από μας. Ευχαριστώ. Κύριε Ριβελίνη. Δεν ξέρω αν ο συμπρόεδρος έχει τίποτα άλλο να πει. Ε, αν δεν έχει τελειώνει η συνεδρίαση, στην επόμενη, η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 13 ε, Ιουλίου μεταξύ 3 και 4 η ώρα, ίδια ώρα δηλαδή. Θα σταματήσουμε τώρα μέχρι τις 4 ε, και 4 και μετά θα αρχίσουμε τις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Όσοι δεν, ε, δεν τους αφορά αυτή η συνεδρίαση μπορούν να αποχωρήσουν. Το επόμενο σημείο που θα συζητήσουμε θα είναι η απαλλαγή του Συμβουλίου. α.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

Λοιπόν, συνεχίζουμε, συνάδελφοι, τη συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Ελέγχου Προϋπολογισμών. Ε, απαλλαγή για το Συμβούλιο. Τώρα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα συνεχίσουμε Έχουμε τον κύριο Κέσλε από τη Γενική Διεύθυνση. Η κυρία Κρέσλε είναι εδώ ως εισηγήτρια. Ο κύριος Ριβελίνη δεν έχει πολύ χρόνο γιατί θα πρέπει να πάει στην Επιτροπή Αλίας και στο τριμερή διάλογο, που θα δώσω το λόγο στον κύριο Ριβελίνη για να μας πει τι, πού βρίσκονται τα πράγματα. Για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι, θα συναντήσουμε, θα συνεδριάσουν οι συντονιστές, θα επιστρέψει ο κύριο Ριβελίνη και στις 6 παρατέταρτο θα συζητήσουμε με το Συμβούλιο το θέμα αυτό. Κύριε Ριβελίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να πάρω ε, μέρος στον τριμερή διάλογο για την αλία. Και επομένως, μετά από αυτήν την παρέμβαση, θα απουσιάσω και θα επανέλθω για την ανταλλαγή απόψεων με τους σκιώδεις εισηγητές. Λοιπόν, θα ήθελα με τη σημερινή συζήτηση καταρχάς να υπενθυμίσω ποια είναι η κατάσταση για το φάκελο, για το θέμα του Συμβουλίου, ούτω ώστε να εξάγουμε κάποια περάσματα για την ε, στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Μετά την παρουσίαση του ερωτηματολογίου στο Συμβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου του 2010 και την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης στις 28 Φεβρουαρίου, ο, το πρόεδρο του, ο πρόεδρος του ελεκτικού συνεδρίου έλαβε ε, μία επιστολή ε, από τον πρόεδρο του Συμβουλίου ε, για την απαλλαγή ε, του 2010 με τα εξή έγγραφα. Τον τελικό προπολογισμό του 2009 με τους παθητικούς και ενεργητικούς λογαριασμούς που αφορούν την εκτέλεση του προπολογισμού. Ένα έγγραφο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύο. Την έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες και ένα δημόσιο έγγραφο που έχει ήδη δημοσιευθεί στο, στην ιστοσελίδα και επομένως υπάρχει στη διάθεση όλων. Τρίτον, την ε, περίληψη του, των εσωτερικών ελέγχων του 2009, που όπως και το έγγραφο για τις χρηματοδοτικές ε, δραστηριότητες υπήρχε και αυτό ήδη. Οι απαντήσεις τώρα στο ερωτηματολόγιο που προτείναμε δεν είναι σε καμία... Α, δεν τις λάβαμε ποτέ, καταρχάς. Στις 2 Μαρτίου του 2011 το ΚΟΡΕΠΕΡ ενέκρινε ένα πρωτόκολλο προθέσεων που χρησιμεύει ως νέα βάση για τις σχέσεις Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την διαδικασία απαλλαγής. Παρά το μνημόνιο, μπορούμε να το θεωρήσουμε ως ε, βήμα προς τα εμπρό σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση του Συμβουλίου, γιατί ξεχωρίζει την ετήσια διαδικασία απαλλαγής από τη διαδικασία του προϋπολογισμού. Παρ' όλα αυτά το Συμβούλιο ζητάει την πλήρη αμοιβαιότητα μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου στις 3 Μαρτίου, ως ε, συντονιστής, έλαβε γνώση του μνημονίου και των εγγράφων που παρουσιάστηκαν και στην ε, συμφωνία θεωρούν ότι δεν είναι επαρκή, επαρκή τα έγγραφα για να δοθεί η απαλλαγή. Στις 21 Μαρτίου, στην επόμενη συνεδρίαση, ε, κρατήθηκε αυτή η θέση και στις 22 Μαρτίου η Κομισιόν υιοθέτησε την έκθεση που συνέστηνε να αναβάλουμε την απόφαση για την απαλλαγή, η Επιτροπή μάλλον. Μια ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου ακολούθησε και το Κοινοβούλιο πρότεινε διάφορες προσεγγίσεις. Το Συμβούλιο δήλωσε ότι θέλει να ακολουθήσει μια ένα πιο περίπλοκο δρόμο. Στην πραγματικότητα δηλαδή τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας διαθεσμικής και το Κοινοβούλιο δέχτηκε να λάβει υπόψη αυτή την αλλακτική λύση. Μόνο αυτή τη στιγμή η ετήσια διαδικασία του 2009 ολοκληρωθεί. Αυτή η απόφαση ελήφθη στις 31 Μαρτίου συγγνώμη, του 2011. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την απαλλαγή στην Ολομέλεια της 10ης ε, Μαΐου 2011, η Προεδρία του Συμβουλίου μέσω του Υπουργού Μπερξέη κάλεσε τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να διορίσει ε, μια ομάδα διαπραγματευτών για να επιληθεί το πρόβλημα της απαλλαγής του Συμβουλίου. Η ψηφοφορία στην ε, Ολομέλεια με μεγάλη πλειοψηφία ε, αποφάσισε και αυτή να αναβληθεί απόφαση για την απαλλαγή του Συμβουλίου και υιοθέτησε το ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε. Ο συντονιστής Κοντ στη συνεδρίαση του Ιουνίου του 2011 έλαβε υπόψη την ψηφοφορία της Ολομέλειας και αποφάσισε η Προεδρία του Συμβουλίου να συμμετάσχει στην επόμενη ανταλλαγή απόψεων, στην επόμενη συνεδρία δηλαδή. Στο μεταξύ, η Προεδρία του Συμβουλίου έγραψε στι 2 Ιουνίου του 2011 μία επιστολή στον πρόεδρο τον κ. Μπούζεκ, η οποία αναφερόταν στη συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια και έλεγε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν συζητήσει μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, κυρίω για δύο θέματα, προετοιμασία του προπολογισμού και η διαδικασία τη απαλλαγή και είπε ότι εφόσον δεν υπάρξει τελικά μία συμφωνία, το Συμβούλιο θεωρεί ότι η απαλλαγή έχει δοθεί με βάση το άρθρο 319 της Συνθήκης. Αυτό για να ενημερώσω όλους τους συναδέλφους για τα, τις διαπραγματεύσεις του φακέλου. Θα ήθελα τώρα να φτάσω σε κάποια τεχνικά συμπεράσματα. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο, ε, όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα, θα πρέπει να είναι υπεύθυνο οικονομικά για το δημόσιο χρήμα ε, που του εμπιστευόμαστε, όπως συμβαίνουν και για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να απαντήσει στα ερωτήματα που διατυπώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικά η Επιτροπή μας. Είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάποια ερωτήματα που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο, ε, γιατί είναι πολύ πιο σημαντικά και αφορούν άμεσα το Συμβούλιο από νομική άποψη και από πολιτική άποψη δεν είναι λογικά τα επιχειρήματα του Συμβουλίου το, οποίο διεκδικεί ότι η απαλλαγή της, Επιτροπής καλύπτει, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλύπτει την απαλλαγή και των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων. Οι νομομαθείς του Συμβουλίου ε, πέρα από την ε, καταγράμμα ερμηνεία λένε ότι υπάρχει και μια τελεολογική ερμηνεία. Δηλαδή, ε, προσανατολίζει το κείμενο προς την έννοια. Τελικά δηλαδή, προς την έννοια που θέλει να υπάρξει, που θέλει να επικρατήσει ο νομοθέτης. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Κάθε δαπάνη που γίνεται ε, με βάση το, το δημόσιο χρήμα ε, του πολίτη, δηλαδή που, ξοδεύει ο πολίτης, θα πρέπει να ελέγχεται από τον πολίτη. Άρα από ποιους, από τους ε, εκλεγμένους του. Επίσης, ε, έχουμε εγκρίνει πριν από ένα χρόνο, λιγότερο από ένα χρόνο, τον προϋπολογισμό της εξωτερικής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Και λέμε ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης παρότι είναι ιονή θεσμικό όργανο και αυτό υπόκειται στη διαδικασία απαλλαγή. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώ, αφού είναι ιονή ε, όργανο, ε, δεν καταλαβαίνει το Συμβούλιο πώς ε, υπόκειται στη διαδικασία απαλλαγή του Κοινοβουλίου. Αφού το, αν δέχεται λοιπόν ότι υπόκειται στη διαδικασία απαλλαγή η υπηρεσία εξωτερική δράση τώρα θα πρέπει να υπόκειται στη διαδικασία ελέγχου μέσω τη απαλλαγή από το Κοινοβούλιο και το ίδιο το Συμβούλιο. Και ε, θα πρέπει να κρατήσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου ω αρχή απαλλαγή. Συζητήσαμε λοιπόν επίση τη δυνατότητα τροπολογία του δημοσιονομικού κανονισμού και επομένω δεν θα επεκταθώ. Θέλω να ακούσω τι σκοπεύει να πει το Συμβούλιο στην ε, συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά, για την πλήρη αυτή παρουσίαση που δώσατε. Νομίζω ότι έχετε καλύψει όλα τα ουσιώδη στοιχεία. Υπάρχουν τώρα κάποιοι συνάδελφοι οι θα θέλουν να λάβουν το λόγο. Έχετε ερωτήσεις, προτάσεις ή... Ο κύριος Ότι θέλει το λόγο καταρχήν. Βεβαίω, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή μας και θέλω να επαναλάβω το ερώτημά μου. Δεν ξέρω που έχουμε βρεθεί για το θέμα αυτό. Αν υπάρχει μια νομική μελέτη, αν θα γίνει μια νομική μελέτη για να μας εξηγήσει ποια είναι ακριβώς τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου σε σχέση με όλο αυτό το πλέγμα θεμάτων. Είχα ιτηθεί σε σχέση με αυτή την αίτηση πριν από κάποιο χρονικό διάστημα και μετά φαίνεται ότι είχε εγγραφεί στη μέση διάταξη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού εγώ λυπάμαι βέβαια για αυτές τις ανταλλαγές απόψεων μεταξύ του Συμβουλίου που λέει έχετε το δικαίωμα εδώ, δεν έχετε το δικαίωμα εκεί και κάνει συγκρίσεις με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και επιτρέψτε μου τώρα να ανοίξω μια μικρή παρένθεση σε σχέση με την σκέψη μου. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουμε να επιλύσουμε τις μεγάλες προκλήσεις ενώπιών μας εάν δεν χρησιμοποιήσουμε σωστά την ε, κοινοτική μέθοδο και όχι πότε την κοινοτική μέθοδο και άλλες φορές την ε, διακυβερνητικού χαρακτήρα. Κάποια στιγμή δεν θα ξέρουμε στην πράξη ποιος έχει τον πολιτικό έλεγχο για όλα αυτά τα κονδύλια. Και αν η διαδικασία διακρατική ή ενωσιακή, κοινοτική δηλαδή. Θέλουν πάντα οι πολίτες να υπάρχει έλεγχος εκτελεστικής εξουσίας και γι' αυτό έχουν τα κοινοβούλια. Τα εκτελεστικά όργανα εδώ είναι η Κομισιόν και το Συμβούλιο και αν δεν υπάρξει διαλεύκανση του ποιο ελέγχει ποιον θα έρθουμε και σε σύγκρουση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θέλω να τονίσω επίσης ότι μετά από τις καθυστερήσεις και τις αμφιταλαντεύσεις για όλα αυτά τα θέματα τα πρώτα μηχανίσματα τα οποία βγαίνουν από τον μηχανισμό ε, χρηματοοικονομικής σταθερότητος και εδώ μιλάμε για 700 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν είναι φιστίκια. Εδώ πρόκειται για μια καθαρά διακυβερνητική διαδικασία. Ποιος θα ελέγξει αυτά τα κονδύλια, ξέροντας ότι αυτό πρόκειται για τη ζώνη του ευρώ και μόνο και δεν υπάρχει κοινοβουλευτική διάσταση στη ζώνη του ευρώ, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πρέπει να αναλάβει αυτό τον έλεγχο. Κατά την άποψή μου αυτό θα ήταν σωστό. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυτή την υπερεθνική ε, οντότητα θα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή θα είναι τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αν θεωρούν κάποιε κυβερνήσει ότι μπορούν να κινητοποιήσουν 700 δισεκατομμύρια ευρώ χωρί κοινοβουλευτικό έλεγχο, αυτό είναι πραγματικά ένα σοβαρό πολιτικό σφάλμα. Εγώ συμφωνώ λοιπόν με τον εισηγητή μα ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να υπόκειται σε πολιτικό έλεγχο, θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων και κυριών για το μη έλεγχο ορισμένων κατηγοριών, αυτό το γνωρίζουμε αλλά δεν θα ήθελα να καταλήξουμε σε μια υπερβολική δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά, γιατί αλλιώς θα υπάρξει και η αντίδραση των Εθνικών Κοινοβουλίων. Υπάρχουν άλλε παρατηρήσει ή αντιδράσεις. Φυσικά η αντιδρασεις φυσικα η επιχειρηματολογια σας θα καταγραφεί και νομίζω και η γραμματεία με έχει πληροφορήσω ότι υπάρχουν δυνατότητε για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά, αλλά θα πρέπει καταρχήν να προχωρήσουμε σε μια συζήτηση με τους συντονιστέ για τα θέματα αυτά. Επομένω, καταγράφω τη θέση σας. Θα πρέπει λοιπόν να έρθετε σε επαφή με τον συντονιστή σας για να εγγραφεί το θέμα αυτό στην ημέρηση για διαταξή μα. Έχετε άλλε παρατηρήσει τώρα? Όχι? Κλείσαμε το σημείο αυτό λοιπόν. Είναι μια ιστορία με πολλές εξελίξεις. Θα επανέλθουμε. Θα συναντήσουμε και τον κύριο Μπεξίμ σε λίγο. Έρχομαι τώρα στο επόμενο σημείο. Αλλά βλέπω ότι η κυρία Γκρέσλε, ή μάλλον δεν βλέπω την κυρία Γκρέσλε, δεν είναι παρούσα η κυρία Γκρέσλε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν κάποιο από το ΕΛΚ ή κάποιο συνεργάτη τη κυρία Γκρέσλε θα μπορούσε να την ειδοποιήσει ότι χρειάζεται η παρουσία της και συγχρόνως εγώ χαιρετίζω την παρουσία του κύριου Κεσλέρ που είναι Γενικός Διευθυντής της ΟΛΑΦ χαιρόμαστε για την παρουσία του μεταξύ ημών και ίσως κύριε Γενική Διευθυντά θα μπορέσετε να έρθετε πλησίον μου εξεβονίμων μου Hello. Θα ακούσουμε er eh, λοιπόν την παρουσίαση. Μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε την κυρία Γκρέσσα γιατί δεν έχει νόημα να ξεκινήσουμε μια συζήτηση τη απουσία Ευχαριστώ που ήρθε Σίγκε. Ε, σταμάτησα λίγο την ε, συζήτηση γιατί δεν μπορούμε να συζητήσουμε ε, χωρίς την παρουσία σου. Ο κανονισμός της Όλαφ, η μεταρρύθμιση της Όλαφ λοιπόν. Οι συγκρούσεις, τα προβλήματα με το Κοινοβούλιο. Ο κύριος Κέσλερ είναι εδώ. Έχει μια προσωπική εμπειρία. Θα μας μιλήσει για αυτήν. Μετά τις παρατηρήσεις που παρουσιάσαμε τελευταία φορά, παρουσία του κυρίου Κέσλερ και του κυρίου Σεμέτας, Επομένω, προτείνω να ξεκινήσετε εσεί για να σπάσετε και τον πάγο. Ευχαριστώ. Δεν μπορεί κανείς να είναι παντού ταυτόχρονα, κανείς δεν λυπάται γι' αυτό περισσότερο από μένα. Είχαμε να προετοιμάσουμε στην Σύνοδο του Συμβουλίου και είμαι μέλος ε, για το ΕΛΚ. Ε, ένα εγχείρημα που δεν οδηγεί σε αποτελέσματα. Πάει να γίνει η ευρωπαϊκή συνήθεια. Αποφάσισαν οι συντονιστές μετά τις, σχετικέ μετά τις ε, σχετικές ανακοινώσεις συμφωνήσαμε να γίνει συνάντηση εδώ μαζί σας και όχι μόνο για τη μεταρρύθμιση της Όλαφ αλλά και το ότι η συνέχεια θα δοθεί στην όλα, αυτή θα κάνει από το και πέρα. Επίσης, τι συνέβη, ε, ποια είναι η νομική θέση της Όλαφ, η σκοπιά της ε, για τα πράγματα και πώς θα συνεχίσουμε. Πιστεύω παρόλα αυτά ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε παρακαλώ Πόσο έχει ε, προχωρήσει η εσωτερική διαδικασία αναδιάρθρωσης της Όλαφ, μας ενδιαφέρει αυτό. Λέτε ότι το οι, μισοί που στις, οι ε, πρέπει να εργάζονται στις έρευνες. Πόσο προχώρησε αυτό το πράγμα. Επίσης, με ποιους συνεργάζεστε για να κάνετε εσωτερική μεταρρύθμιση. Γιατί πολλοί δεν συμμετέχουν, είναι στην όλα αλλά δεν συμμετέχουν στη μεταρρύθμιση. Άρα τίθεται ένα θέμα αποδοχής της μεταρρύθμισης από τους εργαζομένους εκεί. Λοιπόν, πώς έχουν προχωρήσει τα πράγματα, πού έφτασαν εν μεταξύ και επίσης ακούμε τρελά πράγματα σε σχέση με το πώς αντέδρασε η όλα ακούμε στο Κοινοβούλιο. Πείτε μας εσύ λοιπόν τις, εσείς τις διαδικασίες, τα κίνητρά σας, γιατί δράσατε όπως εδράσατε. Όλα αυτά είναι ενδιαφέρον να τα ακούσουμε και χαιρόμεθα που είστε εδώ. Ευχαριστώ. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο από τους ευρωβουλευτές. Η κυρία Τσέσκοβα καταρχήν. Υπάρχει άλλος ευρωβουλευτής που θέλει να πάρει το λόγο για, σε αυτή τη φάση της συζήτησης. Και ο κύριος Μπαλτσίτης, κυρία Τσέσκοβα πρώτη και συνεχεί συνεχεία ο κύριος ε, Κέσλερ. Ε, děkuji za Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Έχω μία ερώτηση που αφορά ένα δικό μας πρόβλημα. Διαπιστώνω ότι η Όλαφ πρέπει να συνεργάζεται με τα κρατήματα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Υπάρχει το σύστημα της συλλογής των δεδομένων από τα κρατημέλη από τη μία και από την άλλη αυτό που ανακαλύπτει η Όλαφ το διαβιβάζει στα εθνικά όργανα. Ξέρουμε ότι κάποια κράτη-μέλη συνεργάζονται μια χαρά με την Όλαφ, αλλά κάποια άλλα έχουν προβληματική θα έλεγα συνεργασία. Επομένως η ερώτησή μου είναι η εξής. Πώς αυτή η συνεργασία και σε ποια βάση διενεργείται. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη συνεργασία, να τη βελτιώσουμε. Πώς η μεταρρύθμιση της νομικής βάσης για την καταπολέμηση της απάτης πώς θα προχωρήσει και πώς θα βελτιωθεί η συνεργασία με τα κρατη βλέπω ότι πολλά πράγματα εδώ στη μοίρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτώνται από τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να μου απαντήσετε λοιπόν, τι γίνεται με αυτή την περιβόητη συνεργασία. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας. Ο κ. Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ. Κύριε Γερικέ Διευθυντά, στα πρόσφατα 1,5 χρόνια συζητούσαμε το έργο της Όλαφ και υπήρξαν ορισμένε ανταλλαγέ απόψεων και διάφορε νομοθετικέ προτάσει σχετικά. Θυμόμαστε επίση τη διαδικασία επιλογή για το Γενικό Διευθυντή τη Όλαφ και τα προβλήματα χρονισμού που συν... συνδεόντουσαν με αυτή. Τώρα έχει περάσει μισό χρόνο και βλέπουμε να αναδύονται και πάλι τέτοια προβλήματα και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Έχουμε καταρχήν την πρόσφατη πρόταση της Κομισιόν η οποία προτείνει η διαδικασία συντονισμού να αντικατασταθεί με μια πιο εύκαμπτη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων. Πώς το βλέπετε αυτό το θέμα, μήπως θεωρείτε ότι θα οδηγήσει στην ακαμπτοποίηση των δεσμών μεταξύ της Όλαφ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και πώς βλέπετε τον κανόνα de minimis. Υπάρχουν προβλήματα εδώ με τους ανθρώπινους πόρους και τις διαδικασίες για την αντιμετώπιση ορισμένων υποθέσεων και επίσης ποια είναι η αποψή σας για, τους, για τα θέματα δημοσίων προμηθειών και τους κανόνες που συνδέονται με αυτές τις διαδικασίες γιατί υπάρχουν κάποιες καταχρήσεις, πολλές καταχρήσεις κονδυλίων σε σχέση με τις διαδικασίες δημοσίων προμηθειών. Πώς μπορεί να βελτιωθεί λοιπόν το σύστημα δημοσίων προμηθειών. Και επίσης <clears throat> με ανησυχεί η γνωμοδότηση της Όλαφ σε σχέση με τη συλλογή δεδομένων στα κρατη και η ανταλλαγή δεδομένων στα κρατη και οι αρχές που συνδέονται με τα θέματα αυτά. Εγώ ξέρω ποια είναι η στάση του Ελεκτρικού Συνεδρίου της Eurojust και άλλων ε, ειδικευμένων φορέων πέραν της Όλαφ για τα θέματα αυτά. Ποια είναι η δική σας θέση όμως. Παρακαλώ. Θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση λεπτομεριακού επίπεδου. Αν μπορεί να μου πει λοιπόν ο κύριος Γενικός ποιοι είναι οι βασικοί τομείς μεταρρύθμισης που έχετε εξετάσει μέχρι στιγμή στην Όλαφ και τι παραμένει ακόμα να γίνει. Και παρέχομαι και στο ερώτημα που έθεσε η κυρία Γκρέσλε και αυτό δεν έκπληξε κανένα γιατί τα έχουμε συζητήσει ήδη μεταξύ των συντονιστών. Υπάρχουν διαφορετικές και αποκλίνει, αποκλίνουσες απόψεις για το αν έχει αρμοδιότητα και δικαιοδοσία η Όλαφ σε σχέση με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι πράγματι είναι έτσι. Το ερώτημα όμως είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει η διοικητική δικαιοδοσία της Όλαφ Μπορείτε παραδείγματος χάρη να μπείτε σε χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε άλλους χώρους ε, ε, θεσμικών οργάνων. Τέτοιου είδους θέματα θα ήθελα να μπορείτε να μου τα εξηγήσετε. Ευχαριστώ. Άλλες παρατηρήσεις. Όχι. Κανείς. Κυρία Κέσλερ, έχετε το λόγο. Α, συγγνώμη κυρία Γκρέσλε. Ξέχασα κάτι. Την περασμένη Παρασκευή στο Συμβούλιο έγινε μια συνεδρίαση για τη μεταρρύθμιση της Όλαφ. Υποθέτω ότι θα είσαστε κι εσείς εκεί. Όχι, στείλατε κάποιον. Τέλο πάντων, μας ενδιαφέρει να μάθουμε πώς κρίνεται τη συζήτηση που έγινε εκεί στο Συμβούλιο. Από τον Νοέμβριο του 2008 δεν έχει ενημερωθεί ο φάκελος αυτός από το Συμβούλιο και εμείς δεν έχουμε παραιτηθεί ακόμα από την ελπίδα ότι κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες θα συνεχιστεί κάποτε η συζήτηση αυτή και μας ενδιαφέρει να μας πείτε εσείς πώς το κρίνετε αυτό. Μάλιστα. Ο κύριος Κέσλερ. Θα σας δώσω πιο πολύ χρόνο από τότε που σας ανακρίναμε για να διοριστείτε Γενικός Διευθυντής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ γιατί είναι και πιο, πολύ πιο δύσκολες οι ερωτήσεις τώρα. Δεν το ήξερα από πριν. Ναι, γιατί τώρα παίρνετε περισσότερα λεφτά. Πάντω εσείς μετά με ενημερώσατε για τα προβλήματα. Πάντως αυτή είναι η δουλειά μου πράγματι. Επιτρέψτε μου να χωρίσω τις πολλές ερωτήσεις σας σε τρία κεφάλαια που έχουν ε, σχέση μεταξύ τους αλλά έχουν και διαφορές. Η διαδικασία της μεταρρύθμισης, ε, αυτό που λέω ο εσωτερικός έλεγχος, τι κάνουμε δηλαδή για να ε, αναθεωρήσουμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες και το θέμα της όλα σε σχέση με το Κοινοβούλιο ή αντίστροφα αν κάποιος ε, υπενήχθη μια σύγκρουση. Δεν ξέρω, πάντως είναι ένα ζήτημα που εξακολουθεί να υφίσταται. Ελπίζω στο τέλος να μην ε, υπάρξει κάποια αντίθεση. Είναι ένα θέμα πάντως. Συν κάποιες άλλες παρατηρήσεις και σχόλια από ορισμένους. Τα τρία βασικά πάντως αυτά είναι. Για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού. Ε, ήμουν εδώ στην Επιτροπή και πήρα και το λόγο γιατί εκλήθη να πω τη γνώμη μου για την πρόταση που έκανε η Κομισιόν και είπα ότι η πρόταση εκείνη κατ' εμέ είναι καλή. Και την προσυπογράφω κι εγώ γιατί συμμετείχα επίσης με κάποιο τρόπο περιορισμένο γιατί μόλις είχα φτάσει, αλλά, μόλις είχα αναλάβει, αλλά συμμετείχα και πριν πάω στην Όλαφ Άρχισε ως Γενικός Διευθυντής στα μέσα Φεβρουαρίου και είχε σχεδόν ολοκληρωθεί η πρόταση μέχρι τότε. Πάντως, μου έδωσε τη δυνατότητα η Επιτροπή, ο Ορμόδιος Επίτροπος, να γνωμοδοτήσω κι εγώ προσωπικά και να κάνω κάποιες προτάσεις που όντως ελήφθησαν υπόψη. Γενικά λοιπόν, αν με ρωτάτε για τη γενική μου γνώμη από αυτού, συμφωνώ και νομίζω ότι είναι καλή ενημέρωση, δεν είναι τεράστια μεταρρύθμιση, απλώς γίνεται μια επικαιροποίηση του ε, τωρινού κανονισμού. Τώρα, ε, θα συνεχίσω τα γενικά σχόλια. Ελπίζω ότι ο ένας κανονισμός θα τροποποιηθεί και θα ε, τεθεί σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατό. Αυτό σημαίνει ότι η Όλαφ δεν μπορεί να δουλεύει καλά σε κατάσταση αβεβαιότητας σχετικά με το μέλλον της και το νομικό της πλαίσιο και το ίδιο ισχύει και για τους εταίρους της. Ήδη λοιπόν θέτουμε κάποιους στόχους ώστε να ευθυγραμμιστούμε με το μελλοντικό κανονισμό, παρόλο που δεν ξέρουμε ακόμα τι περιεχόμενο θα έχει. Μπορούμε να εικάσουμε κάποια πράγματα με βάση την πρόταση της Κομισιόν και με βάση τις συνεχιζόμενες συζητήσεις στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Εκφράζω όμως την επιθυμία, δεν μπορώ να ζητήσω τίποτε, Άλλωστε δεν εξαρτάται από μένα ούτε ε, και από το Κοινοβούλιο αποκλειστικά, αλλά εκφράζω την επιθυμία το, στο τέλος αυτής της, το τέλος αυτής της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας να είναι όσο γίνεται πιο γρήγορα για να μπορέσει να λειτουργήσει όπως πρέπει η Όλαφ. Μια δεύτερη γενική, ε, γενικής φύσεως ευχή ή επιθυμία είναι ο κανονισμός να μην μπαίνει σε υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες. Ε, η πρόταση της Επιτροπής είναι πιο λεπτομερής τώρα από εκείνη της του 1991 που ήταν αρκετά γενικόλογη. Ίσως γι' αυτό να παρέμεινε και αμετάβλητη τόσα χρόνια. Βέβαια χρειάζεται ένας βαθμός λεπτομέρειας, ε, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το δικαίωμα της υπεράσπισης, ε, προστασίας δεδομένων. Αυτά είναι θέματα που πριν από 10 χρόνια και παραπάνω δεν ήταν τόσο σημαντικά όσο είναι τώρα βέβαια. Γι' αυτό είναι σωστό. Αυτά τα θέματα τα ρυθμίζει ο κανονισμός. Άλλα όμως, όπως η εσωτερική οργάνωση, αλλά και γενικότερα. Νομίζω ότι καλύτερα είναι να μην μας βαραίνει πολύ με λεπτομέρειες ο κανονισμός. Να αφήνει κάποια θέματα, ας πούμε συμφωνίες ή διαπραγματεύσεις, να τα αφήνει στη διακριτική μας ευκαιρία. Ή οι σχέσεις με τη Eurojust και τη Europol Προσωπικά δεν πιστεύω ότι εκεί χρειάζονται πολλές λεπτομέρειες και νομοθετικές ρυθμίσεις από τον κανονισμό. Άλλωστε και η Eurojust πρόκειται να μεταρρυθμιστεί και μετά τη μεταρρύθμιση της Eurojust ε, τότε θα πρέπει να κάνουμε άλλες μεταρρυθμίσεις κι εμείς. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ένα τρίτο, μια τρίτη γενική παρατήρηση για τον κανονισμό Ίσως το θέμα είναι δύσκολο και πολιτικής φύσεως. Υπάρχει μια τάση, και συμφωνώ με αυτό, να ε, ε, θεωρήσουμε de facto την Όλαφ μια δικαστική αστυνομία η αρχή. Αναφέρομαι εδώ στον κανονισμό για το δικαίωμα της υπεράσπισης και τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων να ζητήσουν ε, πανεξέταση, ενημέρωση κλπ. Συμφωνώ με αυτά και εν μέρη πρέπει να πω ότι η Όλαφ ε, ήδη λειτουργούσε με αυτόν τον κανονισμό. Είναι εσωτερικός κανονισμός αυτός. Και καλό είναι και σε νομοθετικό επίπεδο να ισχύουν παρόμοιες ρυθμίσεις. Από την άλλη όμως πλευρά αν μας πείτε ότι σε πρακτικούς όρους και έτσι νομίζω με το νέο κανονισμό ότι εμείς έχουμε ουσιαστικά το χαρακτήρα ενός εισαγγελέα και έχουμε κάποια νομικά όρια, εντάξει. Αν δούμε την τρίτη πλευρά τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξουσίες που έχει το γραφείο της Όλαφ ή την εγκυρότητα ως αποδεικτικών στοιχείων των πορισμάτων των ερευνών μας βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο όπως το 1999. Μπορεί να υπάρχει λοιπόν μια έλλειψη ισορροπίας στο τέλος εάν δεν είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί ώστε να μας δώσετε όχι εσείς βέβαια το κοινοβούλιο να είναι τέτοιος ο κανονισμός ώστε να θέσει ένα βάρος, όχι ένα βάρος αλλά ένα πλαίσιο που είναι πάρα πολύ λεπτομεριακό και σωστό, ναι, σωστό το λέω η Όλαφ έχει ήδη ένα τέτοιο πλαίσιο σε σχέση με τις εγγύησεις και τα όρια, τα οποία παρενθετικά ουσιαστικά παρατείνουν τη διάρκεια των ερευνών. Με τρόπο συνεχτικό και συνεχή. Στην τέταρτη τώρα πλευρά έχουμε τις ίδιες περιορισμένες εξουσίες που είχαμε πριν από δέκα χρόνια και δεν ξέρω να έχουμε ένα εκατοστό περισσότερο εξουσίας. Εγώ είμαι διατεθειμένος να παραμείνω στα επίπεδα των εξουσιών που μου έχουν δώσει. Αλλά κατανοώ παρόλα αυτά. Αλλά παραδείγματο χάρη, όταν πρόκειται για τα αποτελέσματα τα οποία μπορεί να εγγυηθεί η εφαρμογή αυτού του κανονισμού, όπω έχει να κάνει παραδείγματο χάρη στην περίπτωση των συνεντεύξεων με τους μάρτυρε έχουν την ίδια εγκυρότητα όταν, όπως είχαν τότε που δεν υπήρχαν περιορισμοί, δεν υπήρχαν κανονισμοί, δεν υπήρχαν εγγύησει. Δεν είναι ότι ζητώ για περισσότερες κρουσίες. Μια μεγαλύτερη εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των ερευνών αυτών των τόσο εγγυημένων εξεταστικών διαδικασιών ώστε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα στα οποία αναφερόταν προηγουμένως η κυρία Τσέσκοβα. Θα ήταν ένας τρόπος να επιτύχουμε με μεγαλύτερη οκίτητα τα αποτελέσματα τα οποία ενδιαφέρουν τις εθνικές αρχές. Άλλο ένα σημείο σε σχέση με τον κανονισμό τώρα. Κάποιος δεν θυμάμαι το όνομά του, συγγνώμη. Αναφέρθηκε στο θέμα της ανταλλαγής απόψεων ούτως υπήν μεταξύ διαφόρων φορέων. Είναι το άρθρο 11α στην πρόταση κανονισμού. Ανταλλαγή απόψεων με τα θεσμικά όργανα. Ολάφ κοινοβούλιο, συμβούλιο και κομισιόν. Δεν φοβάμαι. Αντίθετα, νομίζω θα ήταν πολύ χρήσιμο για την Όλαφ, για το Γενικό Διευθυντή της Όλαφ, να έχει ένα διαθρωμένο διάλογο με τους κύριους εμπλεκομένους, εάν μπορώ να σας αποκαλέσω έτσι, με αυτούς με τους οποίους αλληλεπιδρά και διαδράσετε η ΟΛΑΦ, το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Επίσης, η πολιτική de minimis, de γιατί και αυτή αναφέρθηκε σε μια ερώτηση, θα ήταν η πιο σημαντική στο μέλλον της ΟΛΑΦ. Υποστηρίζω λοιπόν απόλυτα μια τέτοια κατεύθυνση βάσει της πρόταση της Κομισιόν. Δεν θα είναι πια μια διαδικασία de minimis. Ο όρος de minimis είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε de minimis στο εσωτερικό μας. Παρ' όλα αυτά θα είναι οι προτεραιότητες που δίνονται στις έρευνες. Η Όλαφ πρέπει να έχει μια προτεραιοποίηση των προτεραιοτήτων της κατά τη διάρκεια των ερευνών της. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και ένα θέμα το οποίο πιστεύω θα έπρεπε σε ενιάυσια βάση να αποτελεί αντικείμενο απόψε, ανταλλαγών απόψεων με τους εμπλεκομένους με τον διαφανέστερο δυνατό τρόπο διότι αυτό θα βοηθήσει και την όλα. Δεν φοβούμε λοιπόν αυτές τις ανταλλαγές απόψεων. Αλλά πρέπει η διατύπωση να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη προσοχή. Δεν είναι ότι η Κομισιόν ή το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο ότι θα μπορούν να πούνε στην Όλαφ τι θα ψάξει, τι δεν θα ψάξει. Αλλιώς μετατρέπουμε την Όλαφ σε ένα πολιτικό βραχείο ενός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν όμως και όπως έχουν οι κανόνες τώρα, εγώ συμφωνώ με την ιδέα ενός διαρθρωμένου διαφανούς διαλόγου μεταξύ της Όλαφ και όλων των κυριωτέρων συνομιλητών της. Προτιμώ βέβαια να υπάρχει ένας κύριος χώρος όπου όλα τα θεσμικά όργανα θα έρχονται σε επαφή με την Όλαφ. Και τέλος, σε σχέση με τον κανονισμό, η κυρία Γκρέσλα με ρώτησε για τη θέση του Συμβουλίου. Δεν είμαι απόλυτα ενήμερος για το τι γίνεται από ό,τι ξέρω σήμερα <clears throat> δημοσιεύτηκε ένα σχέδιο από τις υπηρεσίες του Συμβουλίου και θα πρέπει να υποβληθεί στην ΜΕΑ τις επόμενες μέρες, επομένως φαντάζομαι θα το έχετε στα χέρια σας πολύ σύντομα. Από ό,τι ήκουσα υπάρχουν ένα ή δύο σημεία τα οποία θα μπορούσαν δυνητικά ενδεχομένω, αλλά εδώ θέλω να παραμείνω σε ασφαλέ έδαφο γιατί δεν έχω άμεσε πληροφορίε σχετικά. Άκουσα ότι ίσω ενδεχομένω φαινομενικά υπάρχει και κάποιο θέμα και κάποιο με ρώτησε σχετικά για το θέμα αυτό, ίσως ο κ. Μπαλσίτη. για την ανταλλαγή δεδομένων με τα κράτη-μέλη. Κάποιο με ρώτησε γι' αυτό. Ο κ. της με ρώτησε. Και στο Συμβούλιο συζητούν πάρα πολύ για την ανταλλαγή δεδομένων με τρίτες χώρε. Αν μου επιτρέπετε, βεβαίω θέλω να προσθέσω κάτι που είναι πιο σημαντικό για μένα. Ανταλλαγή δεδομένων με διεθνεί οργανισμού. Ηνωμένα Έθνη, Παγκόσμια Τράπεζα, που είναι φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε πάρα πολύ σε έρευνες γιατί ως οργανισμοί η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται ευρέως με τα Ηνωμένα Έθνη. Όλο ένα και περισσότερο. Πρέπει να ερευνούμε λοιπόν μαζί και με αυτούς. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα λοιπόν. Και το μήνυμά μου είναι ότι η ανταλλαγή δεδομένων είναι ζωτικού χαρακτήρα για μας. Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Όλαφ και των καθομελών με τις διοκτικές και δικαστικές αρχές. Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της ΟΛΑΦ και ερευνητικών σωμάτων παρόμοιων με την Όλαφ σε διεθνείς οργανισμούς όπως παράδειγμα χάρη ο ΟΗΕ και επίσης ακόμα και αν είναι κάπως διαφορετικό το θέμα αυτό ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Όλαφ και τρίτων χωρών δηλαδή των δικαστικών και αστυνομικών αρχών αυτών των τρίτων χωρών, που εκεί μπορεί να μην έχουν αυτές οι χώρες τους ίδιους κανόνες προστασίας δεδομένων που έχουμε στην Ευρώπη. Με τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ελπίζω ότι δεν θα ανακύψουν νέα προβλήματα σε ό,τι αφορά τον κανονισμό. Ξέρω ότι είναι ένα λεπτό θέμα η προστασία δεδομένων εν γέννη, αλλά όταν αντιμετωπίζουμε το θέμα προστασίας δεδομένων δεν θα πρέπει να, ξεχνάμε ότι είμαστε ένας φορέας διερεύνησης και μερικές φορές είναι απαραίτητη ανταλλαγή δεδομένων. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα συναντηθεί με τον ε, υπεύθυνο για την ε, προστασία δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουμε υποστήριξη και εποπτεία από αυτόν, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε στο Συμβούλιο και περιμένουμε τα αποτελέσματα της απόφασης η οποία θα πρέπει να ληφθεί από εσά με μεγάλη προσοχή και ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση θα γίνει εν τη επιγνώση όλων για τη μεγάλη σημασία της ταχείας και ελεύθερης και πλήρους ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ημών με ΙΤΑ και των άλλων ερευνητικών φορέων. Ένα άλλο θέμα είναι η συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Θα απαντήσω και στο συναφές ερώτημα της κυρίας Τσέσκοβα. Ε, Το θέμα είναι κρίσιμο, γιατί δουλεύουμε και στην τελική η απόφαση δεν λαμβάνεται από την Όλαφ, αλλά λαμβάνονται από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή από τα κράτη-μέλη, από τις δικαστικές κυρίως των κρατών μελών. Εμείς απλώς ερευνούμε και απλώς κοινοποιούμε τα αποτελέσματα. Υπάρχει αυτό το εσωτερικό θέμα, η όλα θα πρέπει να εμπλέξει τις εθνικές αρχές το συντομότερο δυνατόν. Είναι θέμα πολιτικής μας. Θα επανέλθω σε αυτό. Τώρα, τα κράτη-μέλη. Ίσως τον κανονισμό θα μπορούσε να υποθεί κάτι, όπως είπα και πριν. Και με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουν και μεγαλύτερη αξία τα αποτελέσματα των ερευνών μας, αλλά το θέμα είναι αρκετά δύσκολο. Και ίσως τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να διορίσουν, να μας υποδείξουν μια εθνική αρχή ως αρχή αναφοράς. Δεν θυμάμαι το άρθρο που υπάρχει στην πρόταση κανονισμού ε, που αναφέρει τα σχετικά αυτά. Με τις νέες χώρες ε, είναι πιο εύκολα τα πράγματα γιατί ήταν υποχρεωμένες να το κάνουν πριν μπουν στην Ένωση. Ενώ με κάποιες από τις παλιές χώρες ε, υπάρχουν προβλήματα γιατί έχουν είτε εθνική νομοθεσία, έχουν προβλήματα, υπάρχει, υπάρχει θέμα με τις ε, αστυνομίες τους, έχουν πολλές αστυνομίες. Υπάρχει ομοσπονδιοποίηση των κρατών αυτών, καλό είναι βέβαια αυτό, αλλά στη δική μας περίπτωση δεν μας βοηθάει αυτή η ομοσπονδιακή δομή. Ε, δεν είναι εύκολο πάντα να υποδειχθεί ένα εθνικό σημείο αναφοράς ή επαφής. Δεν έχουμε ένα και μοναδικό τέτοιο σημείο για κάθε χώρα. Τώρα, για την εσωτερική αναθεώρηση. Μια και δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερους πόρους. Και ας με διαψεύσετε αν δεν τα λέω καλά εδώ. Αλλά φοβάμαι ότι θα μπορέσετε. Και μια και πρέπει να πλουστεύσουμε, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να είναι πιο ταχύες οι έρευνές μας, βασικά χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους, όπως θύμισε η κυρία Κρέσλερ, αλλά και άλλοι. Περισσότεροι, περισσότερους πόρους χρειαζόμαστε λοιπόν για έρευνες. Και μια και δεν μπορούν να αυγατήσουν οι πόροι, η οποία είναι περιορισμένη. Να ξέρω ότι σας υποσχέθηκα, αλλά είχα υπενηχθεί εδώ και μήνες ότι το θέμα δεν είναι απλώς να πολλαπλασιάσουμε τους ανθρώπους που ασχολούνται άμεσα με τις έρευνες. Και αντί να μιλάω για άτομα, εγώ αναφέρομαι σε πόρους καλύτερα, που είναι και χρόνος Δηλαδή να, να αποδεσμεύσουμε τους ερευνητές από περιτές εργασίες και καθήκοντα και επίσης να αποδεσμεύσετε και την Όλαφ από περιτές εργασίες. Αν δεν το κάνουμε αυτό, κάποιος θα παραπονεθεί, ίσως το κοινοβούλιο. Ε, Παραδείγματο χάρη, έχουμε όλε την, ε, όλες τις που πρέπει να υποβάλουμε. Αν δεν τις κάνουμε θα παραπονηθείτε. Αλλαγή λοιπόν των εσωτερικών κανόνων, των ε, εσωτερικών διαδικασιών των ερευνών. Έχουμε πολλές πλεονασματικέ διαδικασίες που πολλαπλασιάστηκαν μέσα στα χρόνια αλλά που δεν έχουν νόημα. Έχουμε παρακολούθηση, Έχουμε περιπτώσεις συντονισμού, έχουμε περιπτώσεις ε, επικουρίας, έχουμε περιπτώσεις έρευνας, περιπτώσεις αξιολόγησης και τις έρευνες αυτές καθεαυτές επιπλέον. Σε όλε τις στατιστικές όπου αναφερόμαστε η όλα, αναφερόμαστε μόνο στις έρευνες μας. Και που είναι το δεν είναι όλες οι υποθέσεις μας και μόνο το τελικό τμήμα των προσπαθειών. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να απλουστευθούν λοιπόν οι εσωτερικέ διαδικασίε για να κερδίσουμε χρόνο. Να έχουν περισσότερο χρόνο οι ερευνητέ για να ασχολούνται με τι πραγματικέ έρευνε. Να υπάρχει επίση και μεγαλύτερη διαφάνεια. Τα δεδομένα που θα έχετε και που εμεί θα φτιάξουμε θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά έτσι. Εσωτερικά θα κάνουμε την εξή διάκριση ανάμεσα σε δύο καθήκοντα, στα δύο καθήκοντα, πραγματικά καθήκοντα της, ό, της όλα. Ε, έρευνες και δημιουργία πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης. Έχουμε δύο γενικές διευθύνσεις που ασχολούνται με έρευνες. Ε, έχουμε τώρα, αλλά θα έχουμε περισσότερο κόσμο σε αυτές τις ε, ε, γενικές ε, διευθύνσεις και θα έχουμε τη Γενική Διεύθυνση τη Διοικητική. Θα έχουμε τρεις τώρα γενικές διευθύνσεις για έρευνες και μία διεύθυνση για την δημιουργία πολιτικής. Και μία διεύθυνση για διοικητικά θέματα. Το θέμα των πληροφοριών και του follow-up με τα οποία ασχολούνται τώρα 100 άτομα θα απλουστευτούν. Θα παρακολουθούμε λοιπόν και τις υποθέσεις και αφού ολοκληρωθεί η έρευνα, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Θα παρακολουθούμε αυτές οι, τις γενικές διευθύνσεις που δαπανούν χρήματα περισσότερο, αλλά εμείς δεν θα λαμβάνουμε αποφάσεις, δεν είναι δουλειά μας αυτή. Δεν μπορούμε να παγώσουμε τους πόρους. Θα κοιτάμε τις παλιές υποθέσεις. Θα βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι και τι θα έπρεπε να κάνουν. Επίσης προσπαθούμε να δούμε παλιές, παλιότατες δικαστικές υποθέσεις ε, της δεκαετίας του 90 σε τι φάση έχουν φτάσει. Υπάρχουν ερευνητέ δηλαδή ή εισαγγελεί οι οποίοι ασχολούνται με παμπάλε υποθέσεις σε κράτη-μέλη που είναι υποθέσεις φαντάσματα. Και τα τελευταία που κάνουμε στην αναθεώρησή μας, δημιουργούμε μια μονάδα, κεντρική μονάδα, όπου φτάνουν όλες οι πληροφορίες τώρα οι πληροφορίε σήμερα τι πώς έχουν τα πράγματα φτάνουν τυχαία και ως από διάφορες ας πούμε ε, από διάφορους ερευνητές ο Γενικός Διευθυντής δεν ενημερώνεται και ότι θα μπορούσε να ενημερώνεται η απόφαση να ανοίξει μια υπόθεση ή να μην ανοίξει μια υπόφαση δεν ε, λαμβάνεται κεντρικά αλλά τυχαία από έναν ερευνητή από μια μονάδα. Με αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται να δημιουργήσουμε πραγματική πολιτική για τις ε, ερευνητικές προτεραιότητες που απαιτεί ο ενωσιακός, η ενωσιακή νομοθεσία. Για να συνοψίσω, γιατί πολύ πιο γρήγορη πολύ πιο απλή εσωτερική διαδικασία για τις έρευνες. Θα αποδεσμεύσουμε πόρους λοιπόν, θα τους δώσουμε στους ερευνητές και θα κερδίσουν χρόνο οι ερευνητές. Θα γίνονται πιο σύντομα οι έρευνες, θα υπάρχει περισσότερος χρο... κόσμος που θα ασχολείται με τις έρευνες στις α, ε, διευθύνσεις που ασχολούνται με τις έρευνες πραγματικά. Θα ασχολούνται με πληροφορίες, με την ε, με το οικονομικό follow-up καλύτερη διάκριση με τα δύο βασικά καθήκοντα της Όλαφ έρευνας και δημιουργία πολιτικής καταπολέμησης απάτης. Μεγαλύτερη διαφάνεια. Τα νούμερα που έχετε για τους εσωτερικούς μας πόρους σε ερευνητικές υποθέσεις θα είναι πολύ πιο σαφή, θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Με αυτή είναι η στόχη της εσωτερικής μας αναθεώρησης. Κάτι που χρειάζεται, οπωσδήποτε. Η κυρία Κρέσλε ότι, αν κατάλαβα καλά, γιατί άλλαζα κανάλια από τα αγγλικά στα γερμανικά, μπας και καταλάβω, Σας απαντώ και εσάς και στο Κοινοβούλιο. Τι γίνεται με το προσωπικό. Όλο το προσωπικό ασχολείται με τις έρευνες. Θα μπορούσα να είχα και με ένα έγγραφο που θα σας έλεγε τι δουλειά έχουμε κάνει. Δεν το κάνω όμως, γιατί θέλω καταρχήν να εμπλακούν όλοι. Πώς θα το κάνω? Πώς θα υπάρξει απόλυτη δημοκρατία μεταξύ αυτών των 500 ανθρώπων. Αυτή η δουλειά δεν μπορεί να την κάνει ένας άνθρωπος. Ούτε μπορώ να κλωνοποιήσω τους ανθρώπους θα κάνουμε μισή ημέρα συνεδριάσεις μεταξύ των τεσσάρων ε, διευθύνσεων και θα κάνουμε συνεδριάσεις μεταξύ των 22 μονάδων. Κάτσε συνάντηση με μία μονάδα κρατάει μισή ημέρα. Τρεις-τέσσερις ώρες. Πολλαπλασιάστε το με 22 μένουν τέσσερις μονάδες που... Ε, είχαν συνεδρίαση για την εσωτερική αναθεώρηση όλη μέρα. Έχουμε και συνεδριάσεις ε, διευθυντών και δύο συνεδριάσεις ε, του μεσαίου διευθυντικού προσωπικού, ημίσιας διάρκειας, μισή μέρα. Νομίζω ότι θα έχουμε έτοιμο ένα πρώτο σχέδιο για την εσωτερική οργάνωση, τις εσωτερικές διαδικασίες και για το νέο χρηματοδοτικό, τη χρηματοδοτική διάταξη, αφού ολοκληρώσουμε όλες τις διαβουλεύσεις ε, τον Ιούλιο και από την επόμενη εβδομάδα θα έρθουμε σε επαφή με την Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, την Εποπτική Επιτροπή. Θα μπορούσα να το στείλω και στο Κοινοβούλιο και μέχρι το τέλος του 2011 θα εφαρμοστεί πραγματικά. Θα υιοθετηθεί και εφαρμοστεί. The last point. Τελευταίο σημείο. Για την υπόθεση εδώ του Κοινοβουλίου με την Όλαφ. Υποθέτω δεν έχω πια και πολύ καιρό. Καταρχάς ελπίζω να μην πρόκειται για σύγκρουση. Παρότι μοιάζει, βρωμάει λίγο σύγκρουση, έτσι, διελκυστίντα, αλλά ακόμα δεν έχει κλείσει η ιστορία και ελπίζω να τα βρούμε. Οποιαδήποτε ανταλλαγή απόψεων θα ήταν ευπρόσδεκτη, όπως η σημερινή αυτή, περιορισμένη που έχουμε σήμερα. Κάποιο με ρώτησε γιατί ξεκίνησε αυτή την έρευνα, επί ποιας βάσεως. Για μένα είναι αυτονόητο. Αυτή η διαθεσμική συμφωνία που υπογράφτηκε το 1999 από την Κομισιόν, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τον πρόεδρο του Συμβουλίου, που λέει ότι η Όλαφ έχει την εντολή να ερευνήσει για το προσωπικό και τα μέλη της Κομισιόν ακόμα κι αν δεν υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα που εμπλέκονται, ακόμα και αν δεν θίγονται τα οικονομικά συμφέροντα, για οποιαδήποτε ουσιαστική παρατυπία. Αυτή η συμφωνία που λέγεται διαθεσμική συμφωνία αναφέρεται και στον κανονισμό 1073, στην αιτιολογική του έκθεση. Και εφαρμοζόταν από το Κοινοβούλιο. Νομίζω το Νοέμβριο του 1999 εφαρμόστηκε. Στο κεφάλαιο που δεν θυμάμαι το νούμερο, το 14, του δικού σα εσωτερικού κανονισμού, εντάχθηκε δηλαδή, στο δικό σα εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, όπου λεγόταν ξεκάθαρα ότι οποιαδήποτε προβληματική συμπεριφορά ακόμη και αν δεν σχετίζεται με τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαπράτεται από μέλη του προσωπικού ή από τα μέλη των θεσμικών οργάνων, θα πρέπει να αναφέρεται και θα πρέπει να ερευνάται από την όλα. Επομένως, εγώ θεωρούσα ότι είναι προφανές. Εγώ, εγώ, η νομική υπηρεσία και η νομική υπηρεσία της Κομισιόν, με την οποία θα σε επαφή. Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Ούτε μία επιλογή είχαμε έπρεπε να ξεκινήσουμε αδειρήτως μία έρευνα για μία δημόσια υπόθεση η οποία δεν εστρέφεται εναντίον ουδενός και μηδενός. Εμείς ερευνώσαμε ένα θέμα, ένα θέμα που δεν δημιουργήσαμε. Το διαβάσαμε στην εφημερίδα. Και είχα μία πρόσκληση από πολλά μέλη του Κοινοβουλίου που ρωτούσαν τι κάνει όλα αυτή την περίπτωση. Όχι, δεν ξεκίνησα όμως γι' αυτό την έρευνα. Το έκανα διότι υπήρχε μια νομική βάση που μας δίνει τη δυνατότητα όχι να διαλέξουμε, αλλά μας υποχρεώνει να το πράξουμε. Ένα διαφορετικό τώρα ερώτημα. Δεν ξέρω αν το έχει ρωτήσει κανείς, αλλά μπορώ να το ρωτήσω και εγώ ίδιος. Και δεν μπορώ να το ρωτήσω. Είναι αν ε, θεωρείτε εσείς σωστό να ερευνάει όλα αυτό το θέμα αυτό. Εσείς μπορείτε να αλλάξετε τους κανόνες και εγώ δεν έχω κάποια προσωπική γνώμη για το θέμα αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που εμείς ερευνούμε θέματα που αφορούν ευρωβουλευτές. Και κανείς δεν είχε διαμαρτυρηθεί στο παρελθόν. και το θέμα της απουσίας ή της δυνητικής απουσίας βλάβης στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ έχω μία διπλή απάντηση. Ναι. Καταρχήν, ποιο είναι το αποτέλεσμα μιας έρευνας. Δεν το ξέρουμε από την αρχή. Πώς μπορούμε να ξέρουμε από την αρχή ότι δεν υπάρχουν χρηματοδημοσιονομικές πτυχές σε αυτήν την περίπτωση. Ξεκινάμε την έρευνα και βλέπουμε. Και δεύτερον, είναι ηλίου φαϊνότερον. Δεν είναι θέμα ερμηνείας. Αναφέρεται σαφώς στη Διαθεσμική Συμφωνία του 1999, του Μαρτίου μάλιστα, εάν δεν με απατάει η μνήμη μου, και στου στους εσωτερικούς διαδικαστικούς κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρεται ότι έχουμε την εντολή να ερευνήσουμε ακόμα και σε περιπτώσεις όπου δεν εμπλέκεται χρηματικό θέμα. Λυπάμαι όμως, αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη, ότι είπα του κύριου Μπούζεκ, απατάστε κύριε Μπούζεκ, κάνετε λάθος και δεν είναι μοναχα δική μου άποψη. Ίσως όμως αυτή η άποψη δεν υποστηρίζεται από όλους. Ο στόχος μας είναι να είμαστε ανεξάρτητοι και γι' αυτό εγώ επομίζομαι τις δικές μου ευθύνες. Νομίζω ότι έχω μια σωστή νομική βάση σε αυτά τα θέματα <clears throat> και ξέρω ότι και η γραπτή θέση που πήρε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου ήταν πολύ διαφορετική από την προηγούμενη. Σε, τρεις, σε δύο εβδομάδες πήρε τρεις διαφορετικές θέσεις και τις έχω έγγραφες. Και την τρίτη φορά διαδήλωσε δημόσια και αν μου επιτρέπετε εγώ το αντιμετώπισα με πολύ ήπιο τρόπο. Δεν ήθελα δεν ήθελα καμία σύγκρουση μαζί του. Αν ήθελα όμως τώρα να δημιουργήσω μία αντιπαράθεση, θα ήταν πολύ εύκολο για μένα να απαντήσω στη δήλωση του κυρίου Μπούζε. Κάτι το οποίο δεν έκανα. Τώρα εντάξει πρέπει να κλείσω, αλλά είμαι στη διαθεσή να απαντήσω ερωτήματα. Eh, eh, Ευχαριστούμε για αυτήν την πολύ ευρεία ενημέρωση που μας κάνατε. Θα πρέπει να διακόψουμε λίγο πριν από τις 5.30 για να έρθουν οι συντονιστές. Η κυρία Γκρέσλε, ευχαριστώ. Δεν θα μιλήσω για τον κανονισμό, για την Όλαφ τον διαρθρωμένο διάλογο τον βλέπουμε διαφορετικά σε σχέση με την Κομισιόν. Λέμε στη Γερμανία, άμα δεν ξέρεις τι να κάνεις, κάνε μια ομάδα εργασίας. Και αυτός ο διαρθρωμένος διάλογος πολύ μου θυμίζει αυτές τις ομάδες εργασίας χωρίς καμία δέσμευση. Σίγουρα θα επανέλθουμε και στην εναλλακτική της Κομισιόν και εσείς θα χαρείτε γιατί στηρίζουμε την Όλαφ πάνω σε αυτό το ζήτημα. Τώρα, ε, Όλαφ και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρόσβαση στο Προεδρείο. Δεν υπάρχει διαφωνία στο Κοινοβούλιο εδώ σχετικά με το θέμα των ερευνών για τα μέλη και τα οικονομικά του συμφέροντα. Εκεί χρειάζεται η όλα. στα, στα γραφεία των μελών. Ε, ό,τι αφορά την πολιτική εντολή και εδώ υπήρχαν κάποιες ε, ε, προτάσεις ε, που δεν είχαν να κάνουν με το θέμα αλλά με το, τη γενικότερη φήμη των βουλευτών αφορούσαν την πολιτική εντολή λοιπόν των βουλευτών και αυτό πρέπει να το δούμε προσεκτικά γιατί δεν ε, είναι δυνατόν να έρχονται κάθε δεύτερη μέρα και να ε, ψάχνουν τους φακέλους που χειρίζομαι εγώ. Πώς θα γίνει λοιπόν, πώς θα συν... αν ας πούμε γίνονται έρευνες σε γραφεία, ε, θα πρέπει να βρούμε πολιτικές λύσεις διαφορετικές από αυτές που κατέδειξε η Όλαφ αν δεν γίνεται διάκριση μεταξύ ε, οικονομικών συμφερόντων και πολιτικής εντολής, είναι ένα λάθος. Ενδεχομένως ε, δεν μπορούμε να έχουμε εμείς λιγότερα δικαιώματα από τον ε, πολίτη. Οι βουλευτές έχουν κάποια δικαιώματα. Το θέμα της ασυλίας επίσης, πώς θα αντιμετωπίζετε εσείς. κάποια στιγμή είχαμε έναν επίτροπο που δεν είναι πλέον επίτροπος και τον κάλεσε στο γιο του ε, κάποιος, ε, από μια ρωσική επιχείρηση. Και μετά είχε, απέκτησε καθεστώς ε, μάλλον ευνοουμένου ε, ε, εταίρου και ενδεχομένως υπήρχαν κάποιοι λόγοι γι' αυτό. Έτσι θα με ενδιαφέρε να δούμε πώς βλέπει τέτοια περιστατικά η Όλαφ. Θα πρέπει να ε, επικεντρωθείτε και να παραθέσετε παρόμοια περιστατικά και αλλού. Ε, κοινοβούλιο, Κομισιόν. Οι αρμοδιότητες της Όλαφ σε βασικούς τομείς των εργασιών μας που δεν έχουν να κάνουν με την οικονομική διάσταση πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν και να εξηγηθούν. Ο κύριος Οντή σύντομα. Μικρόφωνο παρακαλώ κύριε Οντή. Εγώ νομίζω ότι όποιος λέει ότι κάνει λάθος ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου για το ποιος ελέγχει ποιον και ποιος είναι ο κυρίαρχος ή όχι, αν μία ε, ενισχυμένη πλειοψηφία αντίστροφη είναι επαρκής ή όχι. Εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι ποιος είναι αυτός ο οποίος κάνει τους νόμους και ποιος αποφασίζει το, το δίκαιο και ποιος όχι. Τελευταία ευκαιρία για τους συναδέλφους που θέλουν να λάβουν τον λόγο. Κανείς, κανείς πια. Κύριε Κέσλερ, μπορείτε να κλείσετε τη συζήτηση. Έχετε το τελικό λόγο, αν θέλετε. Νομίζω ότι ήταν λάθο αυτά που είπε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου στι δύο αυτέ επιστολές σε σχέση με τι ε, αρμοδιότητέ μα. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτή είναι μια άποψη την οποία την δημοσιοποίησα απαντώντα με επιστολή στον κύριο πρόεδρο. Αυτό δεν στρέφεται κατά τη ε, εξουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε εναντίον του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβουλίο μπορεί να αλλάξει του κανόνε ανα πάσα στιγμή, να ερμηνεύσει του κανόνε διαφορετικά ή οτιδήποτε τέτοιο. εγώ ερμηνεύω τις αρμοδιότητές μου και αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Αυτής, αυτές είναι και, αυτή είναι και η ταπεινή μου γνώμη. Κυρία Γκρέσλε τώρα αναφέρθηκε σε ένα κάπως διαφορετικό θέμα, το οποίο είναι όμως συνδεόμενο με αυτά που λέγαμε. Συμφωνώ μαζί σας. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, <clears throat> το θέμα αυτό το οποίο αναφέρατε. Δεν είναι θέμα της αρμοδιότητάς μας. Είναι θέμα της δικής σας αρμοδιότητας. Είναι στη δική σας εντολή αυτό. Και εγώ υπήρξα στο παρελθόν μέλος του Κοινοβουλίου, γι' αυτό τα καταλαβαίνω όλα αυτά τέλεια. Και συμφωνώ μαζί σας. Έχετε μια εντολή και η εντολή σας δεν θα πρέπει να επηρεάζεται με οποιοδήποτε ή έμεσο, άμεσο ή έμεσο τρόπο. Μεγάλο το θέμα αυτό. Το ρυθμίσαμε το θέμα αυτό. Δεν μπήκα σε όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά πάντα αντιμετωπίσαμε τα θέματα αυτά με αυροφροσύνη. Απευθυνθήκαμε στο Γενικό Γραμματέα όταν υπήρξε αυτή η περίπτωση με το Κοινοβούλιο. Περίμενα μερικές μέρες, ήρθα μονάχα αφού μίλησα με το Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου. Μου είπε δώστε μου χρόνο και δώστε και στον πρώτο χρόνο να πάρει μια θέση και εμείς το κάναμε αυτό και τον πληροφόρησα εκ των προτέρων προσωπικά. Ήρθα τρεις φορές να μιλήσω με τον Γενικό Γραμματέα εκ των προτέρων προτού προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε δράση. Δεν υπήρχε λοιπόν κάτι το απρόπτο, καμία απρόπτη ενέργεια. Από τη δική μας πλευρά λοιπόν υπήρξε απόλυτη διαφάνεια, <clears throat> απόλυτη συνεργασία, απόλυτη καλοσύνη όπως πρέπει να υπάρχει μεταξύ θεσμικών οργάνων. Δεν φτάνει καλοσύνη όμως. ένας από τους τέσσερις βουλευτές του συναδέλφου σας, ο οποίος, ο οποίος ε, δυσφημίστηκε, όπως λέει, από τις, από τις εφημερίδες αυτές, ζήτησε να μας δοθεί πλήρης πρόσβαση στο γραφείο του τη παρουσία του και ήταν έτοιμος να συναντηθεί μαζί μας. Πληροφορήσαμε τον Γενικό Γραμματέα για το θέμα αυτό και μετά πήρε μια διαφορετική γνώμη ο συνάδελφός σας και άλλαξε την απόψή του, αλλά τελικά επέτρεψε να λάβει χώρα αυτή η έρευνα και τον απαλλάξαμε τελείως. Γιατί κάνουμε μια έρευνα. Και το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν ότι δεν βρήκαμε κάποιο πρόβλημα. Ήταν απόλυτα αθώος. Εκεί καταλήξαμε. Και πράγματι ε, έτυχε μια απόλυτα αθέμητης δυσφήμισης από την εφημερίδα. Τώρα, μου στείλανε και κάποιες επιστολές από παλιά μέλη του Κοινοβουλίου που είπαν ότι θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Αλλά άλλα μέλη του Κοινοβουλίου που είχαμε ζητήσει να γίνουν μάρτυρες, να καταθέσουν ως μάρτυρες για τα θέματα αυτά, είχαν αρνηθεί <clears throat> την συνεργασία τους. Αυτό δεν έχει τίποτα να κάνει με την προστασία της εντολής που έχετε από τους εκλογείς σας ως ευρωβουλευτές. Η πρόσβαση στα γραφεία των βουλευτών προβλέπεται από τον κανονισμό και από την διαθεσμική συμφωνία, αλλά συμφωνώ ότι όταν πρόκειται για μέλη του Κοινοβουλίου θα πρέπει να γίνει μέσα στα πρέποντα όρια τα οποία έχουν να κάνουν με την ιδιαίτερη σας εντολή και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Ήταν περιορισμένη λοιπόν η πρόσβασή μας. Και το μέλος αυτό του Κοινοβουλίου ήταν έτοιμο να συνεργαστεί μαζί μας και έχουμε τρόπους να μπούμε στα γραφεία μονάχα για τους απαιτούμενους σκοπούς και όχι για άλλους. Και αυτό έγινε σε κάποιο βαθμό για το αυστριακό αυτό μέλος το οποίο ενεπλέκεται από τις αυστριακές ε, δικαστικές ανακριτικές μαλλοναρχές οι οποίες ήταν πιο παρεμβατικές από ό,τι οι Όλαφ. Βασιλιωτός κάναμε την έρευνα μαζί τους. Μπορούμε λοιπόν να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά θέλω εσείς να ξέρετε ότι οποιαδήποτε απόφαση που μπορείτε να πάρετε και είναι δικαίωμα σας να πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, διότι εσείς είστε νομοθέτες εγώ όχι. Οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να ληφθεί προσεκτικά γιατί μπορεί να έχει αντικτύπους όχι μόνο σε σχέση με το Κοινοβούλιο αλλά και σε σχέση και με την Κομισιόν γιατί αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο όπως και με εσάς την Κομισιόν και τους αποκεντρωμένους φορείς Οπότε αν δεν έχουμε αρμοδιότητα για, το, για εσωτερικές έρευνες στο Κοινοβούλιο, δεν θα έχουμε εσωτερική δυνατότητα εσωτερικής έρευνας σε κανένα άλλο φορέα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ολοκληρώθηκε βέβαια η συζήτηση επί του θέματος εδώ. Ε, ολοκληρώθηκε η σημερινή κουβέντα μόνο. Ευχαριστώ όλους όσους παρενέβησαν. Παρακαλώ όσους δεν θα παρευρεθούν στην συνεδρίαση των συντονιστών να αποχωρήσουν. Διακόπτουμε ένα-δύο λεπτά και θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών.